Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Καθίστε παρακαλώ. Thank you very much. So I can open the... Ωραία, μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα ασχοληθεί με το μέλλον ε, της ε, κοινωνική συνοχής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, εσάς που δείξατε ενδιαφέρον να συμμετάσχετε σε αυτήν την συζήτηση που αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική ε, συνοχή κατά την άποψη της Επιτροπής μας ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλληλεγγύη και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. χρησιμοποιούμε πολύ χρόνο στην ε, Επιτροπή μας έτσι ώστε να δουλέψουμε ε, για το θέμα αυτό της ε, πολιτικής συνοχής. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις τις, οι οποίες αποτελούν βάση και την, της έκθεσης κυρίας Βέστφα, η οποία είναι εδώ και θα σας τα πει μετά. Επίσης, δουλεύουμε ε, αυτή την περίοδο σε μια έκθεση ε, σχετικά με την 7η ε, έκθεση για την πολιτική συνοχής που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε τον εισηγητή, τον κύριο Μάρκο Ζουλό μαζί μας, ο οποίος στο τέλος της συνεδρίασης θα πει δυο λόγια είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε βεβαίως ε, και την άποψη του Συμβουλίου ε, μέσω της προεδρεύουσας χώρας. Να σας ε, υπενθυμίσω ότι αυτή η έκτακτη συνεδρίαση οργανώνεται με στόχο να ακουστούν οι απόψεις σε διαφόρων εμπλεκομένων μερών και βεβαίως να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με ε, τους ενδιαφερόμενους. Ε, θα ευχαριστήσω όλους ε, τους συμμετέχοντες που εκπροσωπούν διάφορους φορείς και όργανα. Έχουμε την ημερήσια διάταξή μας η οποία αποτελείται από δύο κεντρικά ε, τμήματα. Το πρώτο θα ασχοληθεί με την θεσμική προοπτική, ε, θα μιλήσει το Συμβούλιο, η Κομισιόν, η Επιτροπή Περιφερειών, η Οικονομική και, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και θα έχουμε και εμείς μια σύντομη ε, παρουσίαση συγγνώμη, των δικών μας building blocks. Μετά ε, θα έχουμε ένα δεύτερο πάνελ, ένα δεύτερο γύρο, στη διάρκεια του οποίου θα εκφραστούν οι απόψεις των τοπικών περιφερειακών κοινοτήτων και αρχών όσον αφορά το ίδιο θέμα. Θα ακούσουμε επίσης ε, δύο λόγια ε, για την έκθεσή μας και θα την παρουσιάσει ο κύριος Μάρκο Ζουλό. Έτσι λοιπόν ε, θα προχωρήσουμε ε, στη σημερινή μας συνεδρίαση. Ή να μην χάνουμε λοιπόν χρόνο, επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε. Και πρώτος ε, πανελίστας είναι ο κύριος Νικόλα Ντε Μικέλης από, την, από το γραφείο της κυρίας Κορίνα Κρετσού. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Είμαστε πλέον στην τελική φάση της προετοιμασίας έκθεσης της Επιτροπής. Και όπως ήθεστε με τις τελικές φάσεις, είναι μια επικίνδυνη φάση. Πολλά μπορούν να συμβούν και πολλές σημαντικές αποφάσεις μπορούν να ε, ληφθούν στις επόμενες εβδομάδες. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην χάνουμε την εστίασή μας στο θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες που ο επόμενος προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χρηματοδοτήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Τι περιμένετε από εμά και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω επί του συμπίου αυτού, αλλά υπάρχει ένας κεντρικός στόχος που είναι ακριβώς αυτός της βελτίωσης ε, της ζωής ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε? μέσα από προσιτές βασικές υπηρεσίες μέσα από την υποστήριξη της οικονομικής μετατροπής μέσω της καινοτομίας κλπ. Και φυσικά μέσω της υποστήριξης της καινοτομίας, ε, και την ε, βελτίωση των προγραμμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Βεβαίως, ε, πολλά μπορούν να γίνουν καλύτερα και πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν και κάποιες, κάποιες, κάποιοι νέοι τομείς οι οποίοι προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και που θα απαιτήσουν νέες επενδύσεις σε τομείς όπως είναι ο έλεγχος των συνόρων, η ασφάλεια, η άμυνα. Επομένως, η συζήτηση ε, περί του τι πρέπει να γίνει δεν έχει ολοκληρωθεί σίγουρα. Το δεύτερο ερώτημα, και αυτή είναι η σωστή αλληλουχία σκέψης, το δεύτερο ερώτημα λοιπόν είναι με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτές τις προτεραιότητες με εργαλεία όπως ας πούμε το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, εάν τα εργαλεία που έχουμε για την έρευνα ε, είναι τα καλύτερα, προγράμματα όπως ο Έρασμος ε, για την κινητικότητα και την ανταλλαγή φοιτητών σε όλη την Ευρώπη, αν όλα αυτά είναι καλά. Υπάρχουν όμως και κάποια πεδία ε, ε, στα οποία δυσκολευόμαστε να δούμε ε, πρόοδο εάν δεν υπάρξει, δεν υπάρχει μάλλον διαρκής συζήτηση και διάλογος με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και κοινωνίες όπως είναι η συμπερίληψη, όπως είναι η αποφυγή της κοινωνικής περιθωριοποίησης. η συζήτηση για το κατά πόσον χρειαζόμαστε ε, εργαλεία αποκλειστικής αρμοδιότητας ή κοινή διαχείρισης ε, είναι ε, ψευδής συζήτηση και ψευδές ερώτημα. Χρειαζόμαστε και τις δύο περιπτώσεις. Όσον αφορά την συνοχή και την πολιτική συνοχής. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται εδώ είναι γιατί χρειαζόμαστε πολιτική συνοχή. Θα σας εκπλήσει ίσως αυτό που λέω, αλλά ε, πραγματικά ισχύει. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το σημείο αυτό με τρεις τρόπους. Ο πρώτος, και όπως το αποδεικνύει άλλωστε και η έβδομη συζήτηση για τη συνοχή στην Ευρώπη, οι φραγμοί εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα αυξάνονται σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης. είτε πρόκειται για ε, κόχες ε, αδυναμίας σε αρκετά αναπτυγμένες χώρες, ε, είτε μιλάμε για τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται κάπου περιορισμένα ανάμεσα σε χαμηλή ανταγωνιστικότητα και χαμηλό εργατικό δυναμικό και έλλειψη καινοτομίας, είτε είτε ε, αν μιλάμε για το μεγάλο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας ε, που αντιμετωπίζουν ήδη και θα αντιμετωπίζουν για αρκετό, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα ορισμένες περιφέρειες. Το δεύτερο παραπέμπει στα προηγούμενα που ανέφερα καθορίζοντας ε, τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και στην καινοτομία και στις, ε, στην κοινωνική ε, συμπερίληψη και ε, σε διάφορα άλλα στοιχεία, εργασιακά κτλ. θα πρέπει να εξυπηρετούνται οι προτεραιότητες αυτές από τον προϋπολογισμό. Και ο τρόπος ε, είναι να ξεκινήσει κανείς από τις περιφέρειες που το χρειάζονται περισσότερο. Εάν δει κανείς το, ε, το χάρτη της Ευρώπης, διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα καινοτομίας ε, σε όλες τις περιφέρειες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα μείωσης της ανταγωνιστικότητας. Ε, και ε, ακριβώς εκεί έγκυται το μεγάλο ε, πρόβλημα της Ευρώπης που σχετίζεται ακριβώς με τη γεωγραφική διάσταση της πολιτικής. Και το τρίτο στοιχείο είναι περισσότερο πολιτικής φύσεως. Αυτό που ονομάζουμε εμείς την γεωγραφία της δυσαρέσκειας. Τα τελευταία χρόνια συνενούν όλοι ε, όσον αφορά την ε, γεωγραφική διάσταση των, της οικονομικής δυναμικής. Ε, διαβάζω ένα απόσπασμα από έκθεση που παρουσιάστηκε στον Ταβός. Ο οικονομικός πόνος έχει επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες ομάδες και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες. Υπάρχει και μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που λέγεται Places That Don't Matter, περιοχές που δεν μας νοιάζουν, όπου, ε, που δεν έχουν σημασία, που αναφέρουν ακριβώς ότι δεν ε, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε ε, την περιφερειακή εδαφική διάσταση των ανισοτήτων και θα ήθελα εδώ να σας διαβάσω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ 1973 that launched μια έκθεση του 1973 όταν ξεκίνησε το Περιφερειακό Ταμείο που λέει στην ουσία ότι καμία κοινότητα δεν μπορεί να ε, συντηρηθεί και να διατηρηθεί από τη στιγμή που τα μέλη της κοινότητας αμφισβητούν την αποφασιστικότητα ε, της ίδιας της κοινότητας να προοδεύσει. Το λέω αυτό γιατί στην ουσία αυτή είναι η προβληματική που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά χρειαζόμαστε μια ισχυρή ε, πολιτική συνοχή που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Δυο τελευταία λόγια. Ωραία, όλα τι λέμε, όλα είναι καλά στην πολιτική συνοχή, τέλεια και δεν αλλάζουμε τίποτα. Όχι. Θα ήθελα μάλιστα να αναφερθώ σε κάποια ε, στοιχεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το πρώτο αφορά την γεωγραφική ε, κάλυψη της ε, αντίδρασης. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνουν όλοι το, τη σημασία, τη σοβαρότητα αυτού του θέματος. Μπορεί κανείς να πει ότι αν θέλουμε να αποφύγουμε διαχωρισμού στην Ευρώπη, ένας τρόπος είναι να καλυφθεί η, ε, να μειωθεί μάλλον η κάλυψη της ε, πολιτικής συνοχής. Ενώ εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει η πολιτική αυτή να αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύνολο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο, αφορά την εστίαση της πολιτικής. Ε, η πολιτική αυτή θα πρέπει να κάνει ε, τα πάντα, αυτά τα οποία χρηματοδοτούνται τώρα, ε, Υπάρχει μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με την εστίαση της συγχρηματοδότησης σε λιγότερους και πιο σημαντικούς τομείς. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές προσεγγίσεις. Αναφέρομαι κυρίως στη δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά την καινοτομία, ε, της ε, ε, στρατηγικές εφιούς εξειδίκευσης κλπ. Ίσως τώρα θα πρέπει να ανοίξουμε το σύστημα και να αρχίσουμε να διασυνδέουμε, να αρχίσουμε να δημιουργούμε αλυσίδες αξίας κλπ. Τρίτο ζήτημα το οποίο αποτελεί βέβαια και κύριο στοιχείο της συζήτησης στον προϋπολογισμό, είναι η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε ε, να οικοδομήσουμε την αιρεσιμότητα. Πώς δηλαδή θα πρέπει να λειτουργήσει η πολιτική σε διασύνδεση με το ας πούμε ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτή η συζήτηση παραμένει. Υπάρχει συλλογικό ενδιαφέρον ε, για μια τέτοια συζήτηση έτσι ώστε να υπάρχει λογική και να είναι διαχειρίσιμο οποιοδήποτε σύστημα και αν εφαρμοστεί. Και ακούγονται πολλά γύρω από το τραπέζι και θα ακουστούν και σήμερα φαντάζομαι. Τελευταίο είναι πως είναι δυνατόν να επιταχυνθεί λίγο ε, η πολιτική. Βεβαίως γίνεται με μεγάλη προσπάθεια και όσον αφορά τους ελέγχους και τους λογιστικούς ελέγχους, ε, όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα και τα συστήματα και σίγουρα πολλά μπορούν να γίνουν ε, και στις ίδιες τις περιφέρειες ε, των κρατών μελών μέσω ευθυγράμμισης κανόνων κλπ. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ε, η διαδικασία απλούστευσης ε, αποτελούσε πάντα πρόσχημα είτε για να μην γίνει τίποτα είτε για να μπερδευτούν ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Πιστεύω ότι τώρα είμαστε σε μια φάση όπου μπορούμε να δούμε το φως στο τέλος του τούνελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μικέλης. Προσπάθησα να μην ε, επιμείνω στο θέμα του χρόνου, αλλά δυστυχώς είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να σας παρακαλέσω να μην υπερβαίνετε τα 10 λεπτά. Και τα μέλη ε, της Ρέτζη, μάλλον οι συντονιστές θα μιλήσουν για δύο λεπτά και τα μέλη της Ρέτζη για ένα λεπτό, γιατί έχουμε πολλούς ομιλητές. Πρέπει λοιπόν ε, να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο για να τους ακούσουμε όλους. Η κυρία Ελένα Παυλόβα θα μιλήσει τώρα εκπρόσωπο της ε, Προεδρικής, της Βουλγαρικής Προεδρίας και υπουργό. Κυρία Παυλόβα, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Κυρίε και κύριοι, κύριε Μιχαήλοβα, σας ευχαριστώ πολύ που ε, πήρατε αυτή την πρωτοβουλία και μας καλέσατε ως ε, Βουλγαρική Προεδρία να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντική για εμάς Θέλουμε εδώ να συμβάλλουμε και ε, αμερόληπτα και ουσιαστικά όμως αναλύοντας τις επιμέρους ε, γνώμες να ακούσουμε και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και η δική μας ε, να ακουστεί. Είμαστε λοιπόν αμερόληπτος διαμεσολαβητής εδώ και θέλουμε να δώσουμε το έναυσμα για μια ανοιχτή συζήτηση, όχι μόνο για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις και μετά το Brexit, υπάρχει ο κίνδυνος ε, του χαμηλότερου προπολογισμού και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους. Τώρα όμως πρέπει να περάσουμε σε μια πιο πρακτική συζήτηση για τον αντίκτυπο και για όλα τα σημαντικά που ανέφερε ο κύριος Δεμικέλης προηγουμένως. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση ισορροπημένη για τα επόμενα βήματα. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο και το Μάιο θα έχουμε και το προσχέδιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το περιμένουμε. Μέχρι τότε θα θέλαμε να γίνουν διάφορες συζητήσεις. Στις 12 Απριλίου λοιπόν προγραμματίζουμε ένα ειδικό ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τη συνοχή. Να ακούσουμε λοιπόν τις επιμέρους απόψεις και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος. Μερικές παρατηρήσεις ε, που για μένα είναι σημαντικές. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε το επόμενο πι όχι ως ένα εγχείρημα λογιστικής, αλλά μια διαδικασία εντοπισμού συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, και μακροπρόθεσμων και πιο συγκεκριμένων για την κάθε πολιτική. Μετά, όταν έχουμε ιεραρχήσει τις προτεραιότητές μας και έχουμε θέσει τους ε, στόχους μας για τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πλέον να υπεραμεινθούμε της ε, πολιτικής συνοχής είναι το βασικό εργαλείο ενότητας και αλληλεγγύης, που είναι και ο κοινός μας ε, στόχος ε, στην Ευρώπη. Ενότητα και αλληλεγγύη. Θέλουμε να παρέχουμε περισσότερα στους πολίτες μας, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Η Ευρώπη λοιπόν έχει επανέλθει. Ανακτά τις δυνάμεις της και πραγματικά αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε πια ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθο την ευρωπαϊκή προσθεθμένη αξία των επενδύσεων, αλλά πρέπει να αποσαφηνίσουμε και τον ορισμό. Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω. Τρίτον, να υπάρχει σαφής διασύνδεση με τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει και την αρεσιμότητα. Αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση. Ξέρουμε ότι η πολιτική συνοχή ήταν αυτή που βρισκόταν υπό πολύ στενό έλεγχο και τώρα πρέπει να κάνουμε αυτή τη ριζική ε, μεταστροφή από τη συμμόρφωση λοιπόν να περάσουμε στην απόδοση και στα αποτελέσματα. Αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικός άξονας ε, της πολιτικής συνοχής μας. Παράλληλα, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι απαιτείται απλούστευση. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν προσέγγιση και να δούμε τη διασύνδεση μεταξύ πολιτικής και αιρεσιμότητας, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πλήττεται ε, μόνο η πολιτική συνοχή από την αιρεσιμότητα, από τις περικοπές κτλ. Πρέπει αυτό να εφαρμόζεται οριζοντίως. Για την απλούστευση συμφωνούμε γενικά. Πρέπει να έχουμε ένα απλό εγχειρίδιο κανόνων και συνοχή μεταξύ και των ίδιων των πολιτικών. Γιατί μιλούμε για περιφερειακή ανάπτυξη, για κοινωνικά ταμεία, πρέπει όμως να υπάρχει καλύτερη ε, συνεκτικότητα μεταξύ τους και συμπληρωματικότητα με τις άλλες ε, πολιτικές, ασφάλεια, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, γιατί τελικά η πολιτική συνοχή είναι μια ισχυρή επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή είναι μια σημαντική διάσταση στην οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Γιατί θεωρούμε ότι ο τρόπος που σχεδιάζουμε την πολιτική συνοχή είναι ένας δείκτης εμπιστοσύνης ε, προς ε, την Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν μια ισχυρή πολιτική συνοχή ως επενδυτικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε όλες τις νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέξουμε. να έχουμε σαφείς μακροπρόθεσμες ε, προτεραιότητες και όχι μια πολιτική που συνεχώς ε, βουλώνει τρύπες όπου υπάρχουν κρίσεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πολύ συγκεκριμένους ε, στόχους και αποτελέσματα που περιμένουμε. Πρέπει να σταματήσω εδώ, γιατί δεν έχω χρόνο. Σας διαβεβαιώ όμω ότι εμείς ως Βουλγαρική Προεδρία θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αυτή την ε, συζήτηση. Μετά την έκδοση του προσχεδίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το Μάιο, ε, στις 8 Ιουνίου και με τη στήριξη της Προέδρου θα έχουμε μια μεγάλη διάσκεψη όπου θέλουμε να έχουμε τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα της ε, Προεδρίας μας όχι μόνο για το ΠΔΠ, αλλά και για την πολιτική συνοχή μαζί με το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο και να κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση για το προσχέδιο, το ΠΔΠ, να καταλήξουμε στα συμπεράσματα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Ήδη συνεργαζόμαστε με τους Αυστριακούς συναδέλφους για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία μέσα στους επόμενους μήνε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παπλόβα. Σας ευχαριστώ. ευχαριστούμε που τηρήσατε και το χρόνο σας. Με χαρά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μίχαλ Σνάιντερ που είναι ο εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών για τη σημαντική γνωμοδότηση το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς, κυρία Πρόεδρε, και τα μέλη της Επιτροπής ε, ΡΕΓΚΙ, με την οποία είχαμε πολλές συζητήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Όταν το Μάιο του 2017 περάσαμε μια καλή νομοδότηση, αυτό είναι αποτέλεσμα και της δικής σας συμβολής. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, υποθέτω ότι είναι γνωστές, έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Τα σημαντικότερα μόνο θα επαναλάβω. Καταρχήν αυτά που ελέγχθησαν μέχρι τώρα τα προσυπογράφω και εγώ. Η πολιτική συνοχή είναι η πλέον καλά ελεγχόμενη πολιτική της Ένωσης. Σε πολιτικό επίπεδο ελέγχεται, ελέγχεται από τις ελεγκτικές αρχές, αλλά ελέγχεται και από την επιστήμη που την αξιολογεί και οι περισσότεροι θεωρούν ότι στο παρελθόν η πολιτική συνοχή ήταν πολύ επιτυχημένη και οι διαφορές μεταξύ των αναπτυσσομένων περιφερειών μπόρεσαν να μειωθούν χάρη, την τελευταία δεκαετία, χάρη στην πολιτική συνοχής. Αν δεν υπήρχε η πολιτική συνοχής, και αν τα κράτη-μέλη τα τελευταία 25 χρόνια ήταν υπεύθυνα για την περιφερειακή πολιτική, τότε θα είχαμε ένα patchwork από ε, περιφέρειες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Γιατί κάπου θα είχαν γίνει πολλές επενδύσεις, αλλού δεν θα είχαν γίνει καθόλου επενδύσεις, δεν θα υπήρχαν ε, ενιαία κριτήρια για την ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκά κριτήρια ε, τα οποία εφαρμόζουμε. Αυτή ήταν η βάση της γνωμοδότησης στην Επιτροπή Περιφερειών που ψηφίστηκε το Μάιο με μία ψήφο κατά. Δηλαδή αυτά που ψηφίστηκαν είναι η γνώμη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Τα πιο σημαντικά σημεία εν συντομία η πολιτική συνοχή και στο μέλλον θα πρέπει να είναι μια προσφορά για όλες τις περιφέρειες, όχι μόνο λόγω της αποδοχή τη από τα κράτη-μέλη, αλλά και για λόγου αντικειμενικού. Όλες οι περιφέρειες ε, πρέπει να συμμετέχουν και μπορούν να συμμετέχουν. Η αρχιτεκτονική διάρθρωση, δηλαδή ανάλογα με κατηγορίες περιφερειών, έχει καταξιωθεί και θα έπρεπε να συνεχιστεί. Πιστεύουμε ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι καλό για ε, κριτήριο κατάταξης των περιφερειών στις κατηγορίες, όπως και για την κατανομή των πόρων σε κάθε κράτος μέλος, ε, όπου εκεί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι δείκτες. Πιστεύουμε ότι πέρα από αυτό που ήθιστε, θα πρέπει να προσθέσουμε κι άλλα πιο σύγχρονα στοιχεία και δείκτες όπως ε, δημογραφικούς δείκτες. Έτσι λοιπόν αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν ε, ως κριτήρια. Επίσης η εδαφική, η διαπεριφερειακή συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής. Ε, ε, εκεί γίνεται ορατή η ολοκλήρωση και προωθείται η ολοκλήρωση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η εδαφική συνεργασία θα πρέπει να μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον και, μάλιστα να γίνει και πιο φιλόδοξη. Δεν θα μπω σε επιμέρους στόχους. Όλα αυτά στο μέλλον θα είναι βέβαια δυνατά όταν θα υπάρχει και η απαραίτητη χρηματοδότηση που είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούνται. Έχουμε συζητήσει διαμακρών. Επιλέξαμε μία διατύπωση για το αίτημά μας, αν θέλετε, που λέει ότι πιστεύουμε ότι το ποσοστό στο μελλοντικό προϋπολογισμό πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν ε, τολμάμε να πούμε ότι θα πρέπει ο σημερινός όγκος ε, χρηματοδότης να διατηρηθεί. Μιλάμε για ποσοστό ούτω ώστε να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που προανέφερα. Δεν είναι αυθαίρετο αίτημα, είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων με επιστήμονες. Αν πέσουμε κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε αυτό θα επηρεάσει την κρίσιμη μάζα και δεν ε, θα δεν θα μπορούν να λαμβάνονται ούτε με μονομένα μέτρα, αλλά ακόμα περισσότερο όλο το σύστημα θα υπονομευθεί και δεν θα μπορεί να διατηρηθεί έτσι όπως υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρξει άλλη δομή της πολιτικής συνοχής και δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει μεγαλύτερος φόβος στις περιφέρειες από το να αναγκαστούν να ξαναρχίσουν από το μηδέν. Και οι περιφέρειες και οι ε, ε παραλήπτες της βοήθειας ε, το βλέπουν αυτό σαν εφιάλτη. Τώρα έχουμε τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα και εδώ δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό το απορρίπτουμε ως ε, ανεφαντικημένου εν προκειμένου. Τώρα η σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν πάει πολύ καλά, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί καλά. Δεν την απορρίπτωμε, αλλά λέμε ότι πρέπει να βελτιωθεί. Η πολιτική συνοχή, τα επιχειρησιακά προγράμματα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά οι συγκεκριμένες ε, συστάσεις για τα κράτη-μέλη ζουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Εδώ χρειάζεται λοιπόν καλύτερος συντονισμός για περισσότερες συνέργειες. Πιστεύουμε ότι το δυναμικό ε, είναι τεράστιο και δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί. Στις συστάσεις για κάθε χώρα, ειδικέ για κάθε χώρα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της διαρθωτικής πολιτικής που δεν είναι αιτήσια πολιτική, αλλά έχει μακροπρόθεσμο πολιετή Ανατολισμό. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη τώρα. Μετά το δύσκολο, επίκαιρο θέμα, σύνδεση ε, συνοχή, πολιτική συνοχής, ΕΔΕΤ και τήρηση του κράτους δικαίου με συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Εδώ κάναμε μια δύσκολη συζήτηση στην Ολομέλεια, θέλω να είμαι ειλικρινής ε, υπήρχε μεγάλη ένταση και επιθετικότητα θα έλεγα πράγμα σπάνιο σε εμάς και στο τέλος σχηματίστηκε μεγάλη ευρία πλειοψηφία των μελών της Ολομέλειας που είπαν ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται διαρθρωτικά ταμεία ε, για την εφαρμογή του κράτους δικαίου ή για την ε, υποχρέωση, ε, τον πιθαναγκασμό της συνεργασίας για την αλληλεγγύη. Πρέπει να ξεκαθαρίσω τη θέση μας εδώ. Οι φίλοι της πολιτικής συνοχής πάντα αντιμετωπίζουν πιέσεις. Πρέπει να υπερασπιστούν την πολιτική συνοχής, να δώσουν μάχη για αυτή και πάντοτε κάνουν αναφορά στις συνθήκες, λένε ότι αυτή η πολιτική είναι στις συνθήκες και στις συνθήκες αναφέρονται σαφείς στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με τα πολλά χρήματα που διατίθενται. Και λέγεται πάντα ότι για τα, τους στόχους αυτούς χρειαζόμαστε τα κονδύλια. Είναι εσωτερική ε, είναι δηλαδή οι στόχοι εσωτερικοί στην συνοχή. Τώρα, εάν προσθέσουμε και εξωτερικούς στόχους όπως αλληλεγγύη, κράτος δικαίου, τότε η πολιτική συνοχή θα είναι διαφορετική, θα γίνει αυθαίρετη πολιτική, με ε, τιμωρία και ε, έπαινο. Δεν θα πρόκειται μόνο για αυτό που είναι εμείς, θέλουμε να επικεντρωθούμε στους στόχους που ήδη έχουμε επιλέξει. Αν προσθέσουμε και άλλους εξωτερικούς στόχους, τότε θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και δεν θα ξέρουμε ποια ιδέα θα γεννηθεί το επόμενο έτος και ποια το μεθεπόμενο που θα επηρεάσει την κατανομή των κονδυλίων συνοχής. Ε, δεν θα αναφέρω παραδείγματα, μπορεί όμως να υπάρξουν παραδείγματα, να μην μιλάμε για αλληλεγγύη και κράτος δικαίου του χρόνου, αλλά για άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή που είναι ο στόχος μας. Εδώ λοιπόν ξεκαθαρίσαμε το θέμα στην συντριπτική από τη συντριπτική πλειοψηφία της Ολομέλειας. Ε, τώρα, το εύρος της γραφειοκρατίας και εδώ συμφωνούμε εμείς οι εκπρόσωποι των περιφερειών, των τοπικών αρχών, δεν, ε, ξέρετε ε, τι πρόβλημα δημιουργείται με τις μεγάλες διατάξεις και την καθημερινή τους εφαρμογή. Ε, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η, αυτή η γραφειοκρατία. Ε, πρέπει να κάνουμε πολλές απλουστεύσεις για να είναι αποτελεσματικότερη η πολιτική. Τελευταία παρατήρηση με το μάτι στο ρολόι. Από το Δεκέμβρη υπάρχει το Task Force για την επικουρικότητα την συνέστησε ο Κλοντ Γιούγκερ και ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς το, την παρουσίασε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στο task force αυτό και είναι κρίμα, λείπει η συμβολή του Κοινοβουλίου. Είπαμε λοιπόν πού μπορεί να ε, επικεντρωθούμε στις πολιτικές μας και εδώ μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της επικουρικότητας ε, πολλές προτάσεις για να μειώσουμε, να πλουστεύσουμε κανόνες και να έχουμε μια εδαφική προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει τα κατώτερα επίπεδα πολιτικής για την επίτευξη της, ε, των στόχων της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Βανίρσελ από το Τμήμα Οικονομικής και Πολιτικής ε, Συνοχής από την Ευρωπαϊκή, από το χειρονικό... 10 minutes. Why does the EC... E Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εμείς ζητούμε λοιπόν, λέει ο κύριος Βανίρσελ, ισχυρή συνοχή, και ισχυρή πολιτική συνοχής γιατί στις πόλεις και στις περιφέρειες δημιουργείται η ανάπτυξη και δημιουργούνται οι θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα αυτή συζήτηση αφορά συζήτηση επί των αρχών και όχι για τα χρήματα δεν μιλάμε για μια λογιστική άσκηση. Μιλάμε για την εξέβρεση των προτεραιοτήτων και εδώ η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη τις, τους διαθέσιμους πόρους. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή και αυτό που θα πρέπει να υπερισχύσει είναι ότι εδώ έχουμε την αλληλεγγύη αφενός και την ευθύνη από την άλλη, που θα πρέπει να παραμείνουν άρεκτα συνδεδεμένες. Η περιφερειακή πολιτική εστέφθη από επιτυχία στο παρελθόν. Όμως, είναι σαφές ότι πλέον υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ χωρών και μεταξύ περιφερειών. Και το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό. Ως Ευρώπη μπορούμε να το επιτρέψουμε. Επομένως, πρωτίστως θα πρέπει σε όλες τις ε, μεμονωμένες πολιτικές, ιδιαίτερος δε στην περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχή, να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Θέλουμε ε, Ευρώπη νικητών, και επομένως και των άλλων που θα είναι η Ευρώπη των χαμένων ή θέλουμε επί τη βάση των ευρωπαϊκών αξιών μια Ευρώπη η οποία θα δημιουργεί περίπου ίδιες ίσες προϋποθέσεις για όλους συμπεριλαμβανομένων και των ε, ε, περιοχών ε, που βρίσκονται σε απομονωμένες περιφέρειες και απομονωμένες χώρες. Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή που μου είναι ιδιαίτερος προσφυγής, προσφυλής και στις εκθέσεις τις οποίες, και τις γνωμοδοτήσεις τις οποίες ε, εκπονούμε ε, για τη συνοχή, για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, στις περιφέρειες. Το επαναλαμβάνουμε αυτό. Πιστεύω πραγματικά ότι θα επιβιώσουμε μονάχα εάν προκύψει μια ισχυρή πολιτική συνοχής και σύγκλησης. Η Γερμανία και οι κάτω χώρες κερδίζουν ας πούμε τον αγώνα, ε, είναι πρώτες και η Βουλγαρία και κάποιες άλλες χώρες ε, πάνε πολύ χειρότερα και μένουν πίσω. Υπάρχει φυγή εγκεφάλων, το ξέρουμε, από τη Νότια Ιταλία στη Βόρεια Ιταλία ε, ας πούμε και από νότιες χώρες σε βόρειες. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορούμε να το δεχτούμε συνεχίζοντας την διαδικασία την διαδικασία ψηφιοποίησης, στην ουσία αυτό, αυτή η διάσταση θα ενισχυθεί και δεν θα, δεν θα απαλληφθεί. Επομένως προκύπτει αυτό το ερώτημα, τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Και οι πλουσιότερες χώρες θα πρέπει να θέσουν το ερώτημα αυτό θα πρέπει να προκύψει μία ισχυρή κοινή τάση και σε αυτήν, κατά αυτήν την έννοια η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχή παίζουν εξαιρετικά μεγάλο ρόλο. Και βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχή προσθέτει κάτι στις πολιτικές οι οποίες έχουν λάβει χώρα μέχρι τώρα αν έχουμε ας πούμε, πολιτική μεταφορών, πολιτική καινοτομίας, πολιτική ενέργειας, ποια μπορεί να, ποιο μπορεί να είναι το προστιθέμενο στοιχείο, η προστιθέμενη αξία από άποψη ε, πολιτικής συνοχής ή περιφερειακής πολιτικής. Το πρόβλημα είναι ότι στο παρελθόν είχαμε κάποια χρήματα, τα μοιράζαμε στις περιφέρειες, αλλά μέναμε κατά κάποιο τρόπο ε, ε κλεισμένοι μέσα σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και δράσης θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να σταματήσει και θα πρέπει ε, πλέον να υπάρχει διασύνδεση με άλλες πολιτικές. Το είπε και ο κύριος Δεμικέλης. Θα πρέπει να γίνονται συνδυαστικές πολιτικές και βεβαίως και αλλαγή νοοτροπίας στην Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο και αλλαγή νοοτροπίας και σκέψης και σε πολλές περιφέρειες επίσης οι κυβερνήσεις, οι τοπικές περιφερειακές αρχές, οι αρχές της περιφέρειας θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας ο καθένας στον κόσμο και ότι όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι δράσεις, όλοι οι παράγοντες, όλες οι ομάδες οι οποίες εργάζονται. Ε, το άλλωστε είναι και το σημαντικό στοιχείο της συμπερίληψης της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες αυτές. Και κάτι άλλο. η πόλωση ανάμεσα, διαφοροποίηση ανάμεσα σε αστικές περιοχές και περιοχές της υπαίθρου. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, υπάρχει αυτή η διάσταση και δεν είναι καλή. Δέστε λίγο τη Γερμανία. Όταν η Ανατολική Γερμανία ε, έπρεπε να ενσωματωθεί στην ε, ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, έγινε μια, μια μάχη ανάμεσα στους Γερμανούς και τους Δυτικογερμανούς, τα δύο αυτά κομμάτια ας πούμε, της Γερμανίας, αλλά ξεπεράστηκε. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας και να πούμε ότι μονάχα ε, μια συγκλίνουσα πορεία ε, είναι αυτή η οποία μπορεί να δημιουργήσει ε, μία όχι ομόσπονδη κρατική δομή, αλλά μία ομόσπονδη ας πούμε αντιμετώπιση της Ευρώπης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ ή της Κίνας. Πρέπει όλες οι δυνάμεις να ενωθούν ε, και η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχή μπορεί να βοηθήσει κατά την έννοια αυτή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στα κράτη-μέλη η συνεργασία ως παράγον επιτυχίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Of, ε, Um, um, η ιδέα της ε, συγχρηματοδότησης ε, είναι εξαιρετικά χρήσιμη ε, βάσει των όσων είπα μέχρι τώρα. Ο ε, ιδιωτικός τομέας βοηθάει σε όλες τις διαδικασίες και είναι μακρόθωρος. Ε, δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει τόσα πολλά επιτεύγματα χωρίς τη, τον, τη βοήθεια, τη συμβολή του ε, ιδιωτικού τομέα. Ε, επίσης να σας πω ότι εγώ βλέπω εξαιρετικά θετικά το εξάμεινο. Εγώ ήμουν επικεφαλής της Επιτροπής για την Ευρώπη 2020 ε, ε, στην ΕΟΚΕ και μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές το εξάμεινο. Μπορεί να είναι ένα πολύ επιτυχημένο εργαλείο, αλλά, όπως είπε και ο κύριος Δεμικέλης, μονάχα εάν έχει ε, προσεγγίσεις μακροπρόθεσμες. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βέστφαλ, η συγγήτρια της Επιτροπής μας για τα building blocks ε, για την πολιτική συνοχή μετά το 2020. Παρακαλώ, κύριε Βέστφαλ. Ähm, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω ότι την πολιτική συνοχής ε, τη βλέπω να κινδυνεύει στο μέλλον. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή προχώρησαν με, έκθεση πρωτοβουλίας και είπαμε θέλουμε να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα για τα δομοστοιχεία της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, διότι ε, όχι μόνο με την πρώτη ματιά αλλά και με τη δεύτερη ματιά πιστεύομαι ότι πρέπει να δώσουμε μάχη ώστε η πολιτική συνοχής ε, να προστατευτεί, γιατί ε, διατρέχει κίνδυνο. Μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, ενδεχομένως 12 με 13 δις ευρώ ε, λιγότερα θα μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Όμως τα καθήκοντα στο μέλλον αυξάνονται. Άρα λοιπόν οι ανάγκες για τον προϋπολογισμό είναι πολύ μεγάλες και τα διαρθρωτικά ταμεία είναι που θα βοηθήσουν γιατί πρικοδοτούνται οικονομικά και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πολύ που η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζονται τόσο καλά όχι μόνο εν προκειμένου ε, με βάση αυτές τις ε, εκθέσεις, ε, αλλά και σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας και ο γοητευτικός Γιώσεφ είναι από τις ανατολικές περιφέρειες, εγώ από τις δυτικές και παρόλα αυτά μπορούμε να συνεργαζόμεθα άριστα πρέπει να το λέμε ξανά και ξανά. Τα... Να δούμε τα διαρθρωτικά ταμεία τι ε, προσφέρουν. Δημιουργούν θέσεις εργασίας και αντιμετωπίζουν το τεράστιο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι επενδύσεις στην και η στην έρευνα. Δεν υπάρχει τίποτε πιο απαραίτητο από τις επενδύσεις στην έρευνα σήμερα, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη θέση της Ευρώπης στην έρευνα οι υποδομές σε κάποιες περιφέρειες μπορεί να μην είναι πολύ καλές, αλλά υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Επίσης, τα διασυνοριακά προγράμματα. Ή έχουμε το, την απασχόληση που θα δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες διαπιστώνω συχνά ότι δυστυχώς ε, δεν ε, ασχολούνται όλοι ως, ε, όσοι θα έπρεπε με τα θέματα αυτά. Γι' αυτό ε, τονίζομαι στο Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει αυτή η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση να διατηρηθεί. Η πολιτική συνοχή είναι κάτι παραπάνω από κινητήρια δύναμη για την απασχόληση. Είναι και αλληλεγγύη στην πράξη. Η διαρθρωτική πολιτική είναι ο συνδετικός κρίκος που ε, συνέχει όλες τις πολιτικές. Από τη μία πλευρά ε, ε, ωφελούνται οι κάτοικοι των πόλεων αλλά και των αγροτικών περιοχών των περιφερειών. Η Ευρώπη τι μπορεί να κάνει για μας. Δεν είναι τίποτα αφηρημένο η Ευρώπη. Η Ευρώπη με τα διαρθρωτικά ταμεία ε, μπορεί να γίνει ορατή και ε, ελκυστική. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά για να τονίσουμε την, ε, ε τα θετικά σημεία της Ευρώπης Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την συνέχιση αυτής της πολιτικής. Είναι πολύ καλό διότι ο συνάδελφος Σουλό στην έκθεσή του θα ε, αναφερθεί και στην έκθεση πρωτοβουλίας και σε αυτά τα δομικά στοιχεία. Στην έκθεση ε, βάλαμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, εκεί όπου τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Όσο καλή και να είναι η γενική, γενικά η πολιτική συνοχής, τόσο περισσότερες ανάγκες για βελτίωση έχει. Το είπαμε ήδη αρκετές φορές. Ε, αρχίζουμε με τη γραφειοκρατία. Προφανώς ε, ένα σωρό έντυπα θα πρέπει να συμπληρώνονται, αλλά δεν πρέπει να ε, ε, ε τρομοκρατούμε ε, τους ετούντες ε, σε σημείο τέτοιο ώστε να μην ε, πιάνουν στα χέρια τους τα έγγραφα αυτά και τις αιτήσει. Επίσης δεν θα πρέπει να φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν για τυχόν λάθη. Εμείς θέλουμε μια αντιστροφή αυτής της πολιτικής. Οι άνθρωποι, οι ετούντες συγκεκριμένα, και οι διοικήσεις θα πρέπει να πούν ναι στην Ευρώπη. Οι διοικήσεις θα πρέπει να πούν ναι στις ε, ε, αιτήσει. Ε, δεν θα πρέπει να δρουν τιμωρητικά. Χρειάζονται γι' αυτό απλοί κανόνες και πιο ευέλικτοι κανόνες πάνω απ' όλα. Εμείς και οι περιφέρειες θα πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε σε νέες προκλήσεις. Διότι ίσως το 2024 να είναι τελείως διαφορετικές οι προκλήσεις από τις σημερινές και τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να μπορούν και να αντιδρούν σε αυτές το μέλλον. Γι' αυτό ζητούμε στην έκθεση μια απλή, έναν απλό αναπρογραμματισμό. Θέλουμε ένα λεγόμενο αποθεματικό που ανάλογα με τις ανάγκες θα μπορεί να αξιοποιείται με τρόπο ευέλικτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν να αντιδρούν οι περιφέρειες επιτόπου. Αυτή η ευελιξία αυτού του είδους είναι σημαντική, αναμφίβολα, αλλά δεν αντικαθιστά με κανένα τρόπο τη θεματική συγκέντρωση. Η πολιτική που άρχισε το 2013 είναι καλή και πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον, αλλά δεν, ε, παρόλα αυτά ευελιξία χρειάζεται. Ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό και το ανέφερα είναι η ορατότητα. Θα πρέπει να συζητήσουμε ε, πού βρίσκονται τα ε, πού πάνε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ανακαίνιση κτηρίων, εξυγίανση ε, κτηρίων, κατασκευή μετρό, όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητούμε πολύ συγκεκριμένα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε μια ε, σύγχρονη ε, μη γραφειοκρατική πολιτική συνοχής, μια πολιτική συνοχής και ίσως αυτό δεν το κατανοούν όλοι, αλλά το είπε και η Επιτροπή Περιφερειών, μια ε, πολιτική συνοχή για όλες τις περιφέρειες. Προφανώς υπάρχουν περιφέρειες που χρειάζονται περισσότερα, αλλά υπάρχουν και οι ε, περιοχές υπομετάβαση και πιο αδύναμες. Και ε, ακριβώς εκεί πρέπει να δώσουμε μάχη. Και οι πλούσιες, ε, οι πιο υγιείς περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται λιγότερο από τις πτωχές, αλλά οι κατηγορίες πρέπει να διατηρηθούν και στο μέλλον. Θέλουμε η πολιτική συνοχής να γίνεται για ανθρώπους, για ανθρώπους που ζουν στις πόλεις και θυμάμαι την αντιπαράθεση στο θεματολόγιο για τις πόλεις, ε, όπως και για ανθρώπους που ζουν στο, στην Ήπεθρο. Οι προκλήσεις είναι διαφορετικές στις πόλεις από τις στην Ήπεθρο, αλλά εμείς ε, έχουμε καταρτήσει το θεματολόγιο για τις πόλεις και λέμε ότι ε, έτσι θα ε, ε, έχουμε μία Ευρώπη καλύτερη, πιο κατανοητή και ελκυστική για τους πολίτες. Και οι ε, αντιευρωπαίοι έτσι δεν θα μπορούν να ε, τορπιλήσουν τις πολιτικές μας όταν εμείς θα τις έχουμε θωρακίσει. Στο τέλος θα ήθελα να πω ότι η μάχη αξίζει, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, το ξέρετε όπως και εγώ, η μάχη θα έχει ε, δοθεί και κερδιθεί όταν ε, έχουμε στο τέλος την πολιτική συνοχή που επιθυμούμε. Και μια προσωπική παρατήρηση στο τέλος. Ε, χάρηκα πάρα πολύ διότι η Επιτροπή Περιφερειών τάχθηκε υπέρ της αιρεσιμότητας. Και εγώ έτσι το βλέπω γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια, ένα εμπόδιο που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε το πρώτο πάνελ. Να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Όποιος θέλει να πάρει το λόγο θα έχει τη δυνατότητα. Κύριο Σαμαζέ, παρακαλώ. κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, θέλετε να ξεκινήσουμε από τους συντονιστές. Α, μάλιστα. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Δεν ε, είδα την αντίδραση των συντονιστών. Ξεκινούμε λοιπόν από αυτούς. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ακολουθούμε τη δική σας πρόταση στην αρχή της ε, συνεδρίασης. Δεν ξέρω πώς θέλετε ε, να προχωρήσουμε. Να πω δύο πράγματα. Πρώτον, είναι σαν να είμαστε σε μια οικογενειακή γιορτή. Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της πολιτικής συνοχής. Εκτός από μία-δύο παρατηρήσεις, δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούργιο σε σχέση με αυτά που ξέραμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μήπως όμως θα πρέπει να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση με όσους ε, επικρίνουν την πολιτική μας. Γιατί στην αρχή της περίοδου, 14, 15, 16, πόσα κονδύλια δαπανίσαμε τελικά. είναι σαν τον βάτραχο που τον βάζουν την κατσαρόλα, σιγά σιγά ζεσταίνει το νερό και δεν καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι η αδυναμία, όπως είπε και ο κύριος Βανίλσελ, ότι έχουμε το σχέδιο Juncker, έχουμε διάφορα μέσα και εργαλεία, έχουμε το ΕΦΣΙ, έχουμε παγκόσμιο ανταγωνισμό, έχουμε βαλκανοποίηση της Ευρώπης, στον τρόπο σκέψης, στις αξίες, Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τι ακριβώς μπορούμε εμείς να προσφέρουμε, ποια θα είναι τα, τα βέλτιστα αποτελέσματα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε κάπως τη συζήτηση και έτσι να ακούσουμε τις ε, πιο σημαντικές πληροφορίες. Κάτι από αυτές τις ακούσαμε βεβαίως. η Επιτροπή πρέπει να τα αξιολογήσει καλύτερα τα πράγματα, γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Horizon 2020. Είναι σαν να έχουμε μια πανέμορφη μαζεράτη χωρίς ε, τροχούς, που λείπουν μάλλον δύο τροχοί. Ε, οπότε κάπως ε, τσουλάει, αλλά όχι όπως θα μπορούσε να κινηθεί κανονικά. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στην κυκλική οικονομία και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. και στον κοινωνικό πυλώνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βγάλει τον κοινωνικό πυλώνα από τη συνοχή. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί λένε ότι ο κοινωνικό πυλώνα πάει ξεχωριστά. Εγώ σα λέω και το ΕΛΚ σα λέει ότι αυτό είναι το θεμελιώδε σφάλμα τη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν συνδέονται αυτά τα δύο. Αυτό πρέπει να επικρίνουμε λοιπόν και να πούμε ότι αυτό θα ήταν ε, ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος μετά τα 30 χρόνια της ε, πολιτικής συνοχής. Γιατί και με την κοινωνική διάσταση, την ε, θεματική συγκέντρωση και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να τα δούμε από κοινού. Γιατί φτιάχνουμε υποδομές σε μία περιφέρεια. Έχουμε ευφυή εξειδίκευση. Και με αυτό το συνδυασμό της κατάλληλης κατάρτισης, του κατάλληλου προσανατολισμού και της συνεργασίας και σύμπραξης δημοσιο δυτικού τομέα θα έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Και κάτι τελευταίο. Ποια από αυτά τα χρήματα θα πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη για να τα δίνουμε απευθεία σε αυτούς που αποδίδουν περισσότερο. Παίρνουμε δισεκατομμύρια από την πολιτική συνοχή για να τα βάλουμε στον μηχανισμό διευκολύνοντα στην Ευρώπη, συνδέοντα στην Ευρώπη. Και ξέρουμε ότι τελικά τα κρα... υπήρχαν σημαντικά προβλήματα με τα κράτη-μέλη. Και αν συνδεθούν τα κρατη τότε μπορούν να δαπανίσουν τα κονδύλια. Ιδάλω, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα δαπανίσει. Πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Καλή επταετία. Αλλά αυτό που δεν κατανοούν κάποιοι είναι ότι αλλάζουν οι καταστάσεις τρεις φορές μέχρι να ολοκληρωθεί η επταετία. Το τελευταίο για την προβολή και ορατότητα του έργου μας. Πρέπει η Ευρώπη κάπως ε, να αναζωογονήσει ε, την επικοινωνία που έχει. Είναι κάτι που ήδη κάναμε με την πρόταση Omnibus, αλλά ακόμα περισσότερο. Το ΕΛΚ στηρίζει βέβαια την πολιτική συνοχή στο 95 των όσων ακούσαμε. Thank Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπρέσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να βγάλουμε από το τραπέζι το, ε, ε, αυτό που ακούστηκε ότι αυξήθηκαν ε, οι ανισότητες σε, στην περίοδο κρίσης ναι ενδεχομένως αλλά σε μακρόχρονη θεώρηση οπωσδήποτε οι ανισότητες έχουν μειωθεί αρκεί να δει κανείς τα στοιχεία όπως είναι το ΑΕΠ ας πούμε. Δεύτερον, να θυμηθούμε και να πούμε ότι ενιαία αγορά χωρίς ε, πολιτικής συνοχής ε, δεν είναι δυνατόν να υφίσταται γιατί διαφορετικά ε, τότε θα υπήρχαν χώρες οι οποίες θα έμεναν εξαιρετικά πίσω και τότε οι διαστάσεις θα ήταν πραγματικά εξαιρετικά μεγάλες. Δεύτερον, ζήτημα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης συνέβησαν πολλά, τα οποία ενδυναμώνουν την άποψη ε, όλων μας ε, ότι θα πρέπει η πολιτική συνοχής να αφορεί τους πάντες, διότι αφενός η κρίση διέκοψε τη διαδικασία σύγκλησης, επομένως θα πρέπει να ξαναρχίσει αυτή η διαδικασία για την οικονομία, κυρίως δε για τις περιφέρειες, αφετέρου δε ε, προέκυψαν νέες δυσκολίες, τις οποίες και ο κύριος Ντεμικέλης και άλλοι ανέφεραν. Το γεγονός ότι ακόμα και στο εσωτερικό των πιο πλούσιων χωρών ε, και των πιο πλούσιων περιφερειών εξακολουθούν να υπάρχουν κόχες δυσκολίας και ανέχειας, ε, αυτό καταδεικνύει ότι και περιφέρειες ε, είτε ιδιαίτερα περιφερειακές, είτε ορεινές, είτε ιδιαίτερα μικρής δημογραφικής κάλυψης που μίλης ότι αντιπροσωπεύουν το 80% των περιφερειών. Για όλες αυτές τις περιφέρειες θα πρέπει να ε, ε, ε, υπάρχουν πολιτικές εξειδικευμένες παρέμβασης Δεν αναφέρομαι σε εξειδικευμένες πολιτικές, αλλά να ληφθεί υπόψη αυτή η ιδιαίτερη διάσταση εντός της πολιτικής ας πούμε ψηφιοποίησης ή της πολιτικής για το περιβάλλον κτλ. Επίσης, το ζήτημα των ε, ε, περιφερειών που βρίσκονται σε αυτήν την παγίδα ε, ε, του μέσου εισοδήματος. Ε, γνωρίζουμε ότι ε, ο βιομηχανικός τομέας της Ευρώπης έχει πιεστεί ανταγωνιστικά από το εξωτερικό. Μιλάμε για πιέσεις οι οποίες προέρχονται από το κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και γι' αυτό έχουν ληφθεί και μέτρα άλλωστε. Σε αυτές τις περιφέρειες έτσι ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την ρόμη τους χρειαζόμαστε ε, ειδικά κονδύλια. Πολιτικές λοιπόν οι οποίες θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες δυσκολίες και σε συγκεκριμένα προβλήματα που όμως ε, θα συνάδουν με τους γενικότερους στόχους και πολιτικές της Ευρώπης. Τρίτον, το θέμα των απαραίτητων πόρων. Εγώ πιστεύω ότι ειδικά εμείς ε, που είμαστε κατά κάποιο τρόπο ε, η συμμαχία της ε, συνοχής και των περιφερειών όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών. Είναι ε, φυσιολογικό απέναντι στις ε, νέες προκλήσεις και τις νέες αποφάσεις, ας πούμε, ε, για θέματα όπως είναι η πολιτική άμυνας. Για όλα αυτά, λέω, χρειάζονται καινούρια κονδύλια. Ε, έχουμε το ε, πρόγραμμα Juncker το οποίο κινητοποιεί και ε, χρήματα από την ιδιωτική οικονομία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λειτουργήσει η οικονομία και άρα χρειαζόμαστε πόρους. Νέες προκλήσεις, νέες πολιτικές, νέα και νέα κονδύλια. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια μικρή κουβέρτα πότε να την τραβάμε από τη μία μεριά και πότε να την τραβάμε από την άλλη. Από τη στιγμή που έχουμε νέες δεσμεύσεις θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε και νέους πόρους ακόμα καλύτερα εάν οι πόροι αυτοί είναι ήδη. Το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εγώ πιστεύω ότι και εδώ θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τη σύγκληση. Δηλαδή, είναι ορθόν ότι οι πολιτικές ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα έπρεπε να είναι πολιτικές γενικής φύσεως, μακροοικονομικές αν θέλετε, οι οποίες θα παρεμβαίνουν ε, σε παράγοντες ε, που μειώνουν την ανταγωνιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται σε συντονισμό με την πολιτική συνοχή που παρεμβαίνει αυτή η πολιτική συνοχή στις περιφέρειες και στις σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει επομένως ένα συντονισμό. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει να ενταχθεί σε πολιετή πολιτική γιατί έτσι και αλλιώς δεν είναι δυνατόν να παρέμβει κανείς στην ανταγωνιστικότητα μιας χώρας ε, ε, μέσα σε ένα εξάμεινο και να λύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να ενταχθεί ε, σε ένα πολιετές πλαίσιο με επαλήθευση αναέτος του κατά πόσον έχει λειτουργήσει σωστά το συνολικό και το εξειδικευμένο πρόγραμμα γιατί εδώ μιλάμε ας πούμε για δύο πολιτικές οι οποίες από τη φύση τους ε, είναι ε, πολυετής. Ε, δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να σκεφτεί κανείς να προσαρμόζει την πολιτική συνοχής ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για το όχι που είπατε στην μακροαιρεσιμότητα, γιατί αν ε, προκύψει η μακροαιρεσιμότητα θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μονάχα στην πολιτική συνοχή, γιατί ε, βέβαια καλύτερα να μην υπάρχουν. Είναι καλύτερα να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα κινητροδοτούν και όχι πολιτικές οι οποίες θα τιμωρούν. E οι κανόνες είναι σημαντικοί, οι κοινωνικοί κανόνες είναι πολύ σημαντικοί γιατί άπτονται αξιών όπως είναι η δημοκρατία και ξεπερνούν κατά πολύ τα κλασικά οικονομικά θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να τηρείτε το χρονικό περιθώριο όπως είπα και προηγουμένως. Για να πάρουν όλοι οι συνάδελφοι το λόγο. Ο κύριος από την Άλντε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μείνω στα δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητέ. Τρία ερωτήματα προ τον κύριο Ντεμιχέλης. Γιατί είπατε ότι πρώτα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό αφορά τις προτεραιότητες. Ρωτώ λοιπόν, θα υπάρξει κάποια συνολική σφαιρική στρατηγική ε, μέχρι το 2030 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό συνδέεται άρρηκτα και με το ΠΔΠ. Δεν έχω ακούσει κάτι από αυτό, επομένω τι συμβαίνει. Δεύτερον, πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να συνδέσουμε τα συστήματα περιφερειακής ανάπτυξης και ε, να εξελίξουμε τις ε, πολιτικές ευφυής εξειδίκευσης. Όμως, από εκεί και πέρα, έχουμε ε, κονδύλια μόνο για την ε, ανταλλαγή γνώσεων. Οπότε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, θα γίνει αυτό με επένδυση, για παράδειγμα, στις υποδομές της έρευνας, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. για παράδειγμα, στα επερχόμενα προγράμματα μετά το Interreg Ευρώπη. Και τέλος, γιατί μιλούμε πολύ για την αστική διάσταση των πολιτικών, ποιο θα είναι το μέλλον των αστικών γενοτόμων δράσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια σε αυτό το επιτυχές κατά τη γνώμη μου πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ομαγζή. Και ζητώ συγγνώμη για πριν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα ε, οι αγαπητοί μου ε, συνάδελφοι θα έχουν την ευγένεια να μην με διακόψουν από εδώ και πέρα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που διαφέρει σήμερα. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις κατά τη διάρκεια του 2017 για το μέλλον ε, της πολιτικής συνοχής και τα αποτελέσματα, αποτελέσματα της συζήτησης αυτής συμπεριλαμβάνονται και στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι η έκθεση Westphal. Και στην ε, Επιτροπή Δημοσιονομικών Υποθέσεων έχουμε και την έκθεση το και ολμπραιτ που είναι δύο σημαντικές εκθέσεις για το, μέλλον της, ε, το μελλοντικό ΠΔΠ. Όμως αυτή τη στιγμή ε, βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία, όπου πρέπει να δούμε το μέλλον του προπολογισμού και την αιρεσιμότητα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την κόκκινη ζώνη και τα πάντα θα εξαρτηθούν από αποφάσεις που θα λάβουν άλλοι. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα να σας πω ότι εγώ λυπάμαι λίγο για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει και εμείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είμαστε μάλλον αδύναμοι. Και πιο συγκεκριμένα να το αναφέρω, ε, και ω μέλο της ε, αρμόδια επιτροπή έχουμε δημοσιονομική αδυναμία. Γιατί αν είχαμε ένα πραγματικό κοινοβούλιο που θα μπορούσε να ε, καταρτήσει έναν πραγματικό προπολογισμό και όχι έναν ε, ψευδή, όλα αυτά θα γίνονταν υπό διαφορετικέ συνθήκες και δεν είμαι βέβαιος ότι όλες ε, αυτές οι ευχές που επαναλαμβάνουμε συνέχεια ε, θα μπορέσουν να αντέξουν έναντι της ε, σκληρής στάσης που θα υπάρξει σίγουρα στο Συμβούλιο. Όπου μπορούμε λοιπόν θα πρέπει να τολμήσουμε για να διαφυλάξουμε τα θεμελιώδη και απαραίτητα. Τώρα, μερικά σχόλια επί των όσων άκουσα. Σήμερα υπάρχει κίνδυνος να θυσιάσουμε τις πολιτικές που αποτελούν ε, υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ε, συνθήκες κοινή γεωργική πολιτική, πολιτική συνοχής. Να τα θυσιάσουμε λοιπόν στο βωμό νέων προκλήσεων που συχνά ανταποκρίνονται σε εθνικές αρμοδιότητες και δεν αποτελούν με βάση τις συνθήκες ενωσιακές αρμοδιότητες και ευθύνες. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και τελικά αναδύονται διάφορες αντιφάσεις και αντιθέσεις και ε, κάπως ε, μας φυλακίζουν και μας περιορίζουν. Αν θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, θα πρέπει ε, να μείνουμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και εγώ λέω ότι δεν είμαι ε, υπέρ της πολιτικής ε, ασφαλείας, σε ό,τι αφο... άμυνας μάλλον, στην πολιτική ασφαλεία θα πρέπει η Ευρώπη να συνδράμει, αλλά αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Γνωρίζετε τις θέσεις μου. Το τελευταίο μου σχόλιο, η πολιτική συνοχής. δεν είναι μία νησίδα που δεν έχει καμία σύνδεση με οποιοδήποτε άλλο τομέα πολιτικής. Η πολιτική συνοχή δεν έχει πετύχει όλους τους στόχους της και υπάρχουν ακόμα ανισομέρειες από ό,τι προκύπτει την τελευταία έκθεση. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν ανισομέρειες που προκύπτουν από την ε, παγκόσμια πολιτική οικονομία και ε, αποδυναμώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονό ότι θα πω την απόψή μου, ότι είναι η πολιτική λιτότητας αυτή που ε, αποδυναμώνει τις ε, υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησαμε για την εκπαίδευση, μπορούμε να μιλήσουμε για την υγεία και βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε τους στόχους μας. Γι' αυτό η στήριξη της περιφερειακή πολιτικής στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ήταν μια εξαιρετικά αρνητική απόφαση, όπως και οι ειδικέ αναχώρες συστάσεις. Γι' αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι και θεωρούμε ότι αυτό τελικά σιγά σιγά μας οδηγεί προς τη διολίσθηση ε, από μια πραγματική πολιτική αλληλεγγύης. Τέλος δεν άκουσα στις προτεραιότητε σα τίποτα για την ανέχεια. Γνωρίζουμε ότι δυστυχώ σήμερα η ανέχεια ξαναγίνεται ε, προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδίω στι πλούσιε περιφέρειες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει εκεί προτεραιότητα. Έχω πολλά ακόμα να πω. Όμως, να κλείσω. Σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα η πολιτική μας ομάδα καταρχήν είναι κατά της αιρεσιμότητας. Αλλά εφόσον διατηρείται η μακροοικονομική αιρεσιμότητα από την πλειοψηφία ουσιαστικά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα σήμερα αιρεσιμότητα σε σχέση με την, ε, το σεβασμό του κράτους δικαίου. Γιατί δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι ο σκοπός ε, ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι τελικά η τήρηση των παράλογων αυτών στόχων που τίθενται κάποιες φορές. Ευχαριστώ. Thank you very... πολύ για τους πρασίνους. Ποιος θα μιλήσει από εσάς. Θα μιλήσω στα κροατικά παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος. Η πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα τώρα που συζητούμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit, μετά την έξοδο της Βρετανίας. Πάντα θα υπάρχουν κράτη-μέλη που θα δημιουργούν ανάπτυξη. Όμως, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, ηγέτιδα δύναμη στις τεχνολογίες, στα προστασία του περιβάλλοντος, τα κοινωνικά δικαιώματα. Η κινητήρια δύναμη, η μηχανή αυτή δεν μπορεί να μεταφέρει, να κουβαλάει μόνο λίγα καλά βαγόνια και τα άλλα να αποκοπούν. Πρέπει να βοηθήσουμε τα πιο αδύναμα κράτη να ακολουθήσουν τα πιο αναπτυγμένα. Και το σημαντικότερο είναι το επίπεδο διαβίωσης ε, στα των πολιτών στα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιωθεί. Γιατί σήμερα οι πολίτες ε, κάποιων κρατών μελών, λόγω της φτώχειας που αναφέραμε, φεύγουν από τις πατρίδες τους και πάνε σε πιο πλούσια κράτη και τα πιο αδύναμα κράτη-μέλη ε, υφίστανται μια δημογραφική διάβρωση που πρέπει να ανασταλεί. Και αυτό μας το επιτρέπει η πολιτική συνοχής. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες, το πιο σημαντικό είναι να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και να έχουμε ε, έλεγχο των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για να χρησιμοποιούνται όπως πρέπει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους εισηγητές. Θα φτάσω, θα, θα πω αμέσως ε, τις τελικές μου σκέψεις για να μην ε, μακρηγορήσω. Ο Επίτροπος Ότιγκερ Ήδη αναφέρθηκε στο 10-15% της πολιτικής συνοχής, ε, αλλά στην πραγματικότητα η πολιτική συνοχής ε, αποτελεί την μόνη αναδιανεμητική πολιτική που έχουμε πια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι τελικά κατευθύνονται στην ευρωπαϊκή άμυνα, ε, κονδύλια τα οποία έχουν αφαιρεθεί από την πολιτική συνοχής. Για μία ακόμα φορά λοιπόν ε, βλέπουμε ε, να ε, παίρνουμε χρήματα από τη μία τσέπη για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες πολιτικές. Ενώ μιλάμε για την πολιτική συνοχή, η οποία κατά την άποψή μας θα έπρεπε να παραμείνει πραγματικά ανέγγιχτη. Ε, στην Ολομέλεια ψηφίστηκε ε, μία έκθεση για την καταπολέμηση της φτώχειας με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ε, ένα τέταρτο, 120 εκατομμύρια, ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ευρώπης αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ενώ ε, ε, έχουμε και πολιτικές οι οποίες αφορούν ε, την εγγύηση ελαχίστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της ευρωπαϊκής της φτώχειας. Εμείς συζητούμε ακριβώς να διατηρηθεί ένα αποθηματικό 20% που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους δραστηριότητες, ιδίως δε σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα δεν υπάρχει μια τέτοια ε, αρχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Εμείς πρέπει να πω ε, ε, είμαστε κατά της come fino a sempre fatto, continui adesso la lotta κατά της αρεσιμότητας. Ευτυχώς και κάποιοι συνάδελφοι προηγουμένως ε, ε, αναφέρθηκαν ε, σε αυτό. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βγάλουμε από την να το κεφάλι των περιφερειών που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα πρέπει να πω ότι στα πλαίσια της δέσμης ε, της δημοσιονομικής ε, μεταρρύθμισης που παρουσιάστηκε το Δεκέμβρη από την Κομισιόν, για μία ακόμη φορά βλέπουμε ότι οι κατευθύνσεις ε, οι οποίες αναλαμβάνονται είναι ιδιαίτερως επικίνδυνες, κυρίως δε όσον αφορά την στήριξη των ειδικών προγραμμάτων για την κοινωνική συνοχή, μάλλον για την μεταστροφή των ε, ε, επενδύσεων. Ε, εδώ μιλάμε για 21 δις, για τη χώρα μου θα είναι 2 δις. Και αυτό το Perform Delivery Tool, κατά την άποψή μας, είναι, είναι σημείο το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να επικριθεί. Αυτό το, αυτό το θέμα της απόδοσης δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο ακόμη ομιλητές. Έχετε το λόγο από την Επιτροπή Ρατζιού κύριε Σόλφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο διαπιστώσεις. Καταρχήν, συμφωνώ με αυτά που είπαμε για τη διατήρηση της πολιτικής συνοχής. Δεύτερον, η πολιτική συνοχής θα επιτύχει τους στόχους της μόνο όταν καταφέρει μεταξύ κρατών μελών να αποκαταστήσει μία ισορροπία μειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται κάποια κράτη-μέλη επειδή ωφελούνται από την πολιτική συνοχής να συμβάλλουν ούτως ώστε το κενό αυτό να διευρύνεται. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η πολιτική συνοχής ήταν πολύ σημαντική και για τον εκδημοκρατισμό των δημοσίων επενδύσεων. Υπάρχουν χώρες που αν δεν, αν δεν είχαν πάρει κονδύλια από την πολιτική συνοχής δεν θα ε, έκαναν δημόσιες επενδύσεις δεν θα έδιναν χρήμα δημόσιο στις επενδύσεις. Εκεί λοιπόν όπου στα κράτη που δεν θα γίνονταν δημόσιες επενδύσεις χωρίς πολιτική συνοχή, όπως είπε η συγγήτρια, ε, ωφελούνται και έτσι αποδεικνύεται το όφελος της πολιτικής συνοχής. Θα κάνουμε το παν για να συνεχιστεί η πολιτική αυτή γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μαλέτσης. Τώρα έχουμε τη Βουλγαρική Προεδρία και δίνουμε μεγάλη σημασία στην πολιτική συνοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ρωτώ λοιπόν, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες σε επίπεδο κρατών μελών, διότι Είμαστε πολύ απαιτητικοί όταν μιλάμε για προγραμματισμό, για υλοποίηση, για παρακολούθηση, εκθέσεις. Στον προγραμματισμό λέμε θέλουμε περισσότερες συμπράξεις, δηλαδή αρχές από κάτω προς τα πάνω, εμπλεκόμενοι στα κράτη-μέλη και συντονισμός ε, της πολιτικής με όλες τις άλλες. Αυτά είναι πολύ απαιτητικά και χρονοβόρα πράγματα. Αν αρχίσουμε με τον προγραμματισμό μόνο το 2020, τότε θα έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ την υλοποίηση και στη νέα περίοδο δεν θα καταφέρουμε να έχουμε νωρίς αποτελέσματα ε, στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών. Προφανώς λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε τώρα τον προγραμματισμό και να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα στα κράτη-μέλη για τις προτεραιότητες. Αυτό Συζητήσαμε στην Επιτροπή Ρέτζικ όταν ήρθε και ο Αντιπρόεδρος και ο πρώην συνάδελφος Τόμι Σλάφ είπε ότι ε, δεν ε, είναι εντάξει οι προτεραιότητες για την πολιτική συνοχή και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Χρειάζονται σαφή μηνύματα προς τα κράτη-μέλη, αλλιώς θα καθυστερήσουμε πάλι. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω, γιατί ταυτόχρονα πασχίζομαι με την υλοποίηση αυτή της περίοδου Τώρα μάλιστα αρχίσαμε την ε, υλοποίηση. Πώς θα επιταχύνουμε την ε, ε, υλοποίηση της προηγούμενης περίοδου και να κάνουμε και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη περίοδο. Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση και τα αποτελέσματα για την επόμενη περίοδο. Και αυτά συζητούμε τώρα στα πλαίσια της αιρεσιμότητας. Ποιες θα είναι οι αιρεσιμότητες, θα δημιουργήσουμε εμπόδια ή κίνητρα για την πολιτική συνοχή και την εφαρμογή μέσα από την αιρεσιμότητα. Θα πρέπει να τα δούμε και αυτά. Κάποιοι συνάδελφοι μιλάνε για σύνδεση με την οικονομική πολιτική. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι εδώ, διότι τι είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αφορά τον καθορισμό των καλών οικονομικών πολιτικών, καλών καλού μείγματος πολιτικής για την ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αφορά την αγορά εργασία την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία καλού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, διοικητική ικανότητα δηλαδή αναβαθμισμένη, οπότε πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, πιο συνεκτική, αλλά οι ερασιμότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να δημιουργούν ευκαιρίες και όχι εμπόδια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν ήταν τα σχόλια και οι ερωτήσεις από την Επιτροπή Ρέτζη, κυρίως του συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Και τώρα θα ζητήσω από τους ομιλητές μας να πάρουν το λόγο και να απαντήσουν, να σχολιάσουν ε, τις παρεμβάσεις. Πρώτα οι κυρίες ως συνήθως. Ε, όταν, ε, όταν ζορίζουν τα πράγματα μπαίνουν μπροστά οι κυρίες. Κυρία Παύλοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλιά σας. Να πω πρώτα ότι όντως συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να πολεμήσουμε και να αγωνιστούμε για την πολιτική συνοχή, όχι όμως για την ύπαρξή της, αλλά για τους ε, επιμέρους ε, στόχους. Ήθελα να το πω αυτό. Και όλοι με αφοσίωση εργαζόμαστε γι' αυτό να έχουμε μια συζήτηση ε, για συγκεκριμένους στόχους, ανάλυση των ε, διδαγμάτων που μπορούμε να αντλήσουμε, ανάλυση των νέων προκλήσεων και λήψη αποφάσεων. Τώρα πιο συγκεκριμένα, ναι, αυτή είναι η εθνική μας θέση και από τον ε, αναπληρωτή Πρωθυπουργό κ. Τάνιτ, Το ανέφερε και αυτό σήμερα και το επαναλαμβάνω και εγώ. Αυτό που λείπει είναι ένα μακρόπνο στρατηγικό όραμα για την Ευρώπη έως το 2030. Να αναλύσουμε πού θέλουμε να είμαστε το 2030. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων απέναντι και στις παλαιότερες προκλήσεις, γιατί δυστυχώς ακόμα υπάρχουν ανισότητες μεταξύ χωρών και περιφερειών και μάλιστα κάποιες από αυτές ε, όλο και εντείνονται. Και μετά έχουμε και τις νέες ε, χώρες με νέα προβλήματα και ευρύτερα κλιματική αλλαγή, η πρόκληση της ανέχειας, της ε, κοινωνικής ενσωμάτωσης, ο κοινωνικό πυλώνα που είναι σημαντικός για μας. Να έχουμε μια συνεκτική ε, πολιτική επενδυτική με μια ενιαία δομή. Θέλουμε λοιπόν μια ενιαία πολιτική. Αυτό προτείνουμε και έτσι θέλουμε εμείς ε, να δώσουμε κίνητρα για αυτή τη συζήτηση. Στις 9 Μαρτίου στη Σόφια θα κάνουμε μια σημαντική συζήτηση για το επόμενο ΠΔΠ, το πλαίσιο, του στόχους ε, και ε, τι προτεραιότητε. Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την συνολική εικόνα. Θέλουμε να δούμε ακριβώς τι μορφή θα πάρει το επόμενο ΠΔΠ και μετά θα συνεχίσουμε με την πολιτική συνοχή. Συγκεκριμένη συζήτηση και θα γίνει και για το κοινωνικό ταμείο, για την γεωργική πολιτική, γιατί πρέπει να δούμε όλες τις διαστάσεις. Και μετά κάπως θα πρέπει να τα συνοψίσουμε όλα αυτά σφαιρικά, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα του συνόλου της κατάστασης. για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμιχέλης, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, αυτό για την ε, συνεκτικότητα που ανέφερε και ο κ. Ρόι. Αν υπάρχει μια πολιτική, πολιτική που είναι διατομεακή, αυτή είναι η πολιτική συνοχή, γιατί μας επιτρέπει να συγκεράσουμε διάφορους ε, τομεί. Φτάνει αυτό? Όχι. Σίγουρα πρέπει να δούμε πώς ε, ε, θα διασφαλίσουμε την συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αν δείτε το, τη δέσμη της 6 Δεκεμβρίου, υπάρχει έννοια της εθνικής πλατφόρμας, που είναι ακριβώς ένας τρόπος να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία, το πώς θα συγκεράσουμε όλα αυτά τα επιμέρου στοιχεία, προκειμένου όταν θα έχουμε διάφορες πηγές χρηματοδότησης προς μια περιφέρεια ή χώρα, ε, θα λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Η τρίτη διάσταση είναι αυτή του εξαμήνου. Όλη αυτή η συζήτηση για την διακυβέρνηση αφορά τη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσει και τις επενδύσεις. Αν λέμε ότι τα εγκριτικά ταμεία είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό εργαλείο τη Ευρώπη, δεν μπορούμε να μείνουμε έξω από αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να συμμετάσχουμε. Και αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο να θίξουμε το θέμα που αναφέρατε, ότι πρέπει να είναι αμφίδρομη διαδικασία. Αν θέλουμε να έχουμε λόγο, πρέπει να συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Επομένω, το ζήτημα κατά πόσο η πολιτική συνοχή θα πρέπει να εντάσσεται ή όχι στην ευρύτερη συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση ε, δεν έχει νόημα, γιατί όντω είναι τμήμα τη συζήτηση και θα πρέπει και εμεί ε, ε, να το πάρουμε απόφαση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεύτερον, απορρόφηση. Πολύ σωστά κάνατε και το θίξατε, γιατί είμαστε το 2018, τα πράγματα δεν είναι ιδανικά. Ωστόσο, με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. Το 50% των πόρων της ε, συνοχής, πολιτικής συνοχής έχουν διοχετευθεί ε, σε συγκεκριμένα ε, προγράμματα. Δύο εκατομμύρια έργα έχουμε που ήδη λειτουργούν, 8.000 επιχειρήσεις, πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε στήριξη για, τις, για θέσεις απασχόλησης όλο αυτό βέβαια δεν τα απαραίτητα στις ε, αιτήσει χρηματοδότηση, γιατί αυτό είναι λογιστικό στοιχείο. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την πολιτική και το μέσο, πρέπει να χρησιμοποιούμε ακριβώς τι ίδιε παραμέτρους, γιατί όταν μιλούμε την πολιτική συνοχή, μιλούμε για τις πληρωμές, ενώ όταν εξετάζουμε ευρύτερα πολιτικέ, στρεφόμαστε σε άλλα στοιχεία. Πρέπει λοιπόν σε συγκρίσιμα στοιχεία να βασίζουμε τις περάσματά μας. Το τρίτο αφορά την πληροφόρηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι ακόμα πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχή είναι ποδηλατόδρομοι και πισίνες. Αυτό είναι μια καρικατουρική ε, παρουσίαση του ζητήματος, γιατί εμείς ή μάλλον ε, δικό μα ρόλο είναι να εξηγήσουμε ότι η πολιτική συνοχή δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολύ περισσότερα. Ε, και το παράδειγμα που αναφέρατε είναι εξαιρετικό. Πρέπει κάθε φορά να χρησιμοποιούμε τέτοια παραδείγματα. Παρεπιπτόντως, ακόμα και ο ποδηλατόδρομος είναι σημαντικό και έχει την αξία του αν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερη πολιτικής ε, ενός Δήμου. Από μόνο του δεν φτάνει βέβαια, αλλά ποτέ δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το μεμονωμένο έργο, αλλά ευρύτερα τις στρατηγικές στις οποίες εντάσσεται το καθέργο. Κάτι τελευταίο για τα τρία ερωτήματα που θίξατε. Διάδοχος ε, του, της Ευρώπης 2020. Συνεχίζεται η συζήτηση έχει σχέση και με τους ε, αναπτυξιακούς στόχους ω σημείο αναφορά. Ε, δεν είμαι σίγουρο ότι με τι επόμενε εβδομάδε θα ολοκληρωθεί αυτό ο διάλογο, αλλά κινούμαστε προ αυτήν την κατεύθυνση. Μετά για την καινοτομία. Ο τρόπος, ε, τι λέμε σωστικά, πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης με τους Δήμους και τις περιφέρειες. Αυτά είναι οι στόχοι μα. τι θέλουμε να πετύχουμε και μετά τα κράτη-μέλη, τοπικέ και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να βρουν ε, το ακριβές μείγμα ε, για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Γιατί από πλευρά δημοσίου διαλόγου τον, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι αν θα χρηματοδοτήσουμε ένα μέτρο, ένα ερευνητικό κέντρο ή, ή μια πολιτική. Θέλουμε να δούμε αν θα επιτευχθεί ο στόχος. Και με τη συμμετοχή βέβαια και με τα πανεπιστήμια. Αυτή είναι λοιπόν μια αλλαγή παραδείγματος ε, που έχει ήδη ξεκινήσει στην τρέχουσα πραγματική περίοδο και θα πρέπει να ενισχυθεί για την αστική καινοτόμο δράση. Δεν έχει ληφθεί απόφαση κατά πόσο θα πρέπει ε, να συνεχιστεί στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνολική αστική διάσταση ε, της πολιτικής συνοχής. Στην τρέχουσα περίοδο, λοιπόν, έχει λίγο κατακαιρματιστεί σε διάφορα μέσα. 5% και αστική καινοτόμως δράση, μπορούμε όλα αυτά κάπως να τα συγκεντρώσουμε και να τα εντάξουμε σε μια ε, πιο ισχυρή αστική διάσταση και μετά να δούμε αν απαιτούνται συγκεκριμένε αστικές και ανάτομες δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε και εσείς να πάρετε το λόγο. Μάλιστα. Δύο λόγια από πλευρά μου. Λαμπέρτ, δεν συμφωνώ όταν λες ότι ακολουθούμε την πεπατημένη και ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ διαφορετική ε, ατμόσφαιρα διαπιστώνω, αλλά υπάρχει ένα κλίμα φόβου ότι χάνουμε χρήματα. Και όταν υπάρχει αυτός ο φόβος πρέπει να αναρωτηθούμε, και σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, αν οδεύουμε καλά. Νομίζω ότι ένα από τα κέρια σημεία που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι θα πρέπει να φύγουμε από τη λογική των πυλώνων στην κοινωνική και περιφερειακή πολιτική. Ε, αυτά εντάσσονται σε μια πολύ ευρύτερη στρατηγική. Και όπως ανέφεραν πολλοί ομιλητές προηγουμένως, πρέπει να πρόκειται για ένα συνεκτικό σύνολο που θα φέρει την ανανέωση και αναζωγόνηση της κοινωνίας μας, να ανταποκριθούμε στην αλλαγή παραδείγματος που έτσι και αλλιώς πραγματοποιείται, είτε το θέλουμε είτε όχι, και να διαμορφώσουμε μια νέα βάση για καλύτερο βιτικό επίπεδο και πιο ποιητική εργασία. Η περιφερειακή πολιτική λοιπόν εντάσσεται στη συνθήκη, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ξεχωριστό κεφάλαιο. Αλλά να συνδράμει όλες τις υπόλοιπες πολιτικές. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Η κυρία Μπρέσο λέει όχι με χρήματα όμως ναι, εν μέρη συγχρηματοδότηση με άλλα έργα και συγχρηματοδότηση από τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη. Κύριε Ντεμικέλης, αυτές οι εθνικές πλατφόρμες, θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν. Υπάρχουν και αλλού αντίστοιχες πλατφόρμες, καινοτομία, ψηφιοποίηση και εμείς τα έχουμε αυτά. Μπορούμε να έχουμε μία σειρά εθνικών πλατφορμών, αλλά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μας βοηθάει. Για να βοηθηθούμε πρέπει να βρούμε συμμάχους. Αν μείνουμε μόνοι μας, χάνουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε συμμάχους ε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής για να διαπιστώσουν οι ίδιοι ότι καλώς εκείνους θα κάνει να ε, αν υιοθετήσουν πτυχές της ε, πολιτική συνοχή. Και αυτό ισχύει και για τα κρατημέλη. Όλοι ξέρουμε ότι το ΠΔΠ θα είναι ε, πραγματικό πεδίο μάχη μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ πολιτικών. Αυτό που μετράει είναι η προστιθέμενη αξία. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο εσείς ως ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης μαζί και με τα κόμματα που ε, εκπροσωπείτε να δείτε τι ακριβώς θέλετε να στηρίξετε. Ο Τραμπ εκλέχθηκε από οπισθοδρομικές ε, περιφέρειες μετά από ένα χρόνο τα μοναδικά αποτελέσματα που έχει φέρει είναι να κάνει πιο πλούσιους τους πλούσιους και πιο φτωχούς τους φτωχούς. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Μιλούμε εδώ για τις ευρωπαϊκές αξίες. Οι ευρωπαϊκές αξίες διαφέρουν. Συμφωνώ με τον Λάμπερτ. Δεν γίνεται να βγάλουμε τον κοινωνικό πυλόν από την πολιτική συνοχή. Αυτή είναι η ουσία. Τέλος, για το εξάμεινο. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την χρησιμότητα του εξαμήνου. Πάντα θεωρείται ένα μακροοικονομικό μέσο, αλλά δεν είναι. Αν δείτε τις ειδικέ αναχώρες συστάσεις, υπάρχουν πολλές συστάσεις για την πολιτική καινοτομία, μακροοικονομικές πολιτικές, μικρομεσές επιχειρήσεις, ενεργειακή πολιτική, κλιματική αλλαγή γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για την ε, περιφερειακή πολιτική και τη διαχείρισή της. Ας πούμε, να προτείνουμε και στους άλλους ότι εμείς είμαστε περήφανοι της πολιτικής συνοχής και θα πρέπει να εντάσσεται στο εξάμεινο προκειμένου να διατηρηθεί. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά ήταν πολύ ενθαρρυντικά, η κυρία Βέστιφαλ. Um, πολύ σύντομα. Είναι μεγάλη μου χαρά που κάθομαι δίπλα σου γιατί υπάρχουν ε, πολλές συνέργειες, πολλές ε, φρέσκες ιδέες που προστίθενται ε, και από την Επιτροπή των Περιφερειών. Άλλωστε γι' αυτό φτιάξαμε αυτή την, την έκθεση πρωτοβουλίας για να αντιδράσουμε έγκαιρα ε, βουλευτές που ήταν και στην προηγούμενη θητεία θα θυμούνται πώς αρχίσαμε όλο το πρόγραμμα, όλο τον, ε, τον προγραμματισμό με το γενικό κανονισμό που, ανε, που, οι συνάδελφοι Λάμπερτ και Κρέα ήταν ε, υπεύθυνοι. Όταν τελειώσαμε δεν είχαμε καταλήξει σε... δεν υπήρχε προϋπολογισμός. Γι' αυτό λέμε και γι' αυτό ακούω με χαρά ότι η Βουλγαρική Προεδρία το έχει υπόψη της και θα το προωθήσει. Πρέπει να κινηθούν τα κράτη-μέλη. Θυμίζω αυτό που είπε και η συνάδελφος Αμάτο. Αν ε, κάνουμε περικοπές 10 ε, με 15% αυτό τι σημαίνει συνάδελφοι. Απλώς σημαίνει ότι πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες θα βγουν από την πολιτική συνοχή και τα διαρθρωτικά ταμεία εκτός από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Τι θα γίνει με το αστικό θεματολόγιο που αποφασίσαμε με την πανοκρουσίες και που μας κάνει περήφανους και που τη δεχτήκαμε όλοι. Όλα αυτά που προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσα από εκεί δεν θα γίνουν. Πρόκειται για τους ίδιους πόρους. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν περισσότερα χρήματα στον ενωσιακό προϋπολογισμό. Η Σοσιαλδημοκρατία, και μιλώ για το δικό μου κόμμα, έχει κάνει σαφείς δηλώσεις ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα, γιατί η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης και η αλληλεγγύη είναι που διακυβεύονται. Γι' αυτό Μπορούμε να μιλάμε για προτεραιότητες, για θέματα, θεματική συγκέντρωση, αλλά αν δεν υπάρχουν χρήματα και αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα, τότε η Ευρώπη, όπως είπες, χωρίς να γενικολογείς, αλλά πολύ συγκεκριμένα, τότε ε, θα ε, αποσυναρμολογηθεί ολόκληρη η Ευρώπη και θα έχουν κερδίσει αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη και αυτοί που θέλουν να μην υπάρχει αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Όχι, διάλειμμα δεν προβλέπει. Δεν έχουμε διάλειμμα γιατί δεν θα έχουμε διαφορετικά αρκετό ε, χρόνο. Πραγματικά πρέπει να ε, συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με το επόμενο πάνελ. Είναι ένα πάνελ το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των ενώσεων δήμων και κοινοτήτων και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αναλίζα Μπόνη, η οποία είναι Γενική Γραμματέας της EuroCities. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που καλέσατε τη EuroCities σε αυτήν την ε, συζήτηση. Όπως υπόθηκε, η διαδικασία της πολιτικής συνοχής ήταν πιο δύσκολη αυτή τη φορά από άλλες λόγω του Brexit, λόγω των νέων προτεραιοτήτων, λόγω ε, της ιεραρχήσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ε, λόγω των αιρεσιμοτήτων ε, διαφορετικών και ψευδών αρμοδιοτήτων κτλ. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανοίξουν τα μάτια αυτών που δεν μπορούν να δουν τη διασύνδεση ανάμεσα στη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα ε, για την συνοχή ε, με την συζήτηση που λαμβάνει η χώρα για το μέλλον της Ευρώπης. Σήμερα περισσότερο από ποτέ. Να περιμένουμε λέει ομιλήτρια λίγο για να φύγουν όλοι. Σας διακόπτω λέει η Πρόεδρος. Μπορώ να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, οι οποίοι εγκαταλείπουν την αίθουσα να το πράξουν ησύχως. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε κυρία μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η συζήτηση για την ε, συνοχή να μπει στο κέντρο και σε διασύνδεση με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, γιατί εδώ μιλάμε για αξίες αλλά μιλάμε και για εργαλεία ε, που θα διασφαλίσουν την ενότητα και ε, ποια είναι αυτή η συγκολητική ουσία ε, που διατηρεί ενωμένα τα στοιχεία αυτά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε ήδη ένα κομμάτι. Πώς μπορεί να τα συγκρατήσει μαζί. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η συγκολητική ουσία, αυτή είναι η κόλλα, αν θέλετε, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να παραμείνουν συγκολλημένα κατά κάποιο τρόπο τα προγράμματα και τα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσουμε τώρα από τα βασικά γιατί έτσι πρέπει να ξεκινάμε πάντα και για να διασφαλίσουμε ότι η συζήτηση για την πολιτική συνοχής παραμένει στο επίκεντρο της Ευρώπης. Εάν ανατρέξει κανείς στο λεξικό ε, θα, για να δει τις τρεις αυτές ε, λέξεις θα δει ότι η διασύνδεση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συζήτηση περί αυτού ε, είναι πολύ ε, σαφής. Χρειαζόμαστε ένα ενωτικό σπίτι ε, και η πολιτική συνοχής είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που θα συγκρατήσει ενωμένων τον ευρωπαϊκό οίκο. Όπως είπε και ο κύριος Λάμπερτ, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες Όταν έχουμε μια πολιτική, όπως ας πούμε την πολιτική συνοχής, ε, πρέπει να την υλοποιήσουμε έτσι ώστε να υλοποιηθεί με το πιο δίκαιο και το πιο σωστό τρόπο. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτή είναι και η αδυναμία ε, που αντιμετωπίζουν σήμερα και οι πόλεις. Ε, γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να δουλεύουμε με τις πόλεις, γιατί οι πόλεις είναι σημαντικοί εταίροι σε αυτήν την διαδικασία. Πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην διεύρυνση της πολιτικής συνοχής που θα κάνει την Ευρώπη πιο ε, ε, ισχυρή, μα πολλά πράγματα μπορεί να μην πάνε καλά σε οποιαδήποτε πολιτική η φάση σχεδιασμού είναι ουσιώδου σημασία. Εάν σε αυτή τη φάση ε, τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε δεν πρόκειται να πάνε καλά ούτε μετά. Εάν δεν γίνει λοιπόν μια σωστή διάγνωση στην αρχή και εάν δεν διαμορφωθεί το πρόγραμμα σύμφωνα με αυτή τη διάγνωση, ε, τότε δεν θα ε, προχωρήσει, προχωρήσει σωστά. Εάν η πρώτη φάση, η οποία παίρνει και χρόνο, δεν καθοριστεί σωστά, τότε ε, ε, θα υπάρχει πρόβλημα. Η έλλειψη διαλόγου, η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί ε, πρόβλημα η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ευρωπαϊκό, το εθνικό, το τοπικό, περιφερειακό επίπεδο αποτελεί πρόβλημα. Εάν λυθεί αυτό, τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Ε, στην φάση υλοποίηση τα πράγματα μπορεί να πάνε άσχημα. Εάν ε, δεν υπάρχει ισχυρή ε, ιδιοκτησία των προγραμμάτων, τότε θα υπάρξει αποτυχία. Εάν δεν έχετε σωστή διακυβέρνηση, τότε θα έχετε ακόλουθα και έλλειψη αποτελεσματικότητας. Ε, επομένως τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να ε, λύνονται ε, ένα-ένα και επίσης και η περιπλοκότητα των προγραμμάτων μπορεί να σχετίζεται με το χαμηλό επίπεδο φιλοδοξίας ε, γνωρίζουμε ότι ε, οι πόλεις ε, πρέπει να κάνουν καλύτερες πολιτικές, χρειάζονται μάλλον, είναι απαραίτητες οι πόλεις στη διαμόρφωση των σωστών πολιτικών, γιατί ακούν τον πολίτη, γιατί υλοποιούνται οι πολιτικές επιτόπου, γιατί έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν πραγματικά, γιατί σε αυτό το επίπεδο υπάρχει λογοδοσία, γιατί έχουν την ικανότητα ε, να καινοτομούν, να αντιδρούν σε προβλήματα με διαφορετικό τρόπο συνδημιουργούν με την κοινωνία των πολιτών και με τους πολίτες. Τέλος, οι πολίτες, ε, συγγνώμη, οι πόλεις αποτελούν ε, το απάβγασμα πολλών αρχών Τι ζητούμε λοιπόν ε, έτσι ώστε να βελτιωθεί αυτό το εργαλείο που είναι ε, σημαντικό γιατί αποτελεί τη συγκολητική ουσία για το μέλλον. Ζητούμε καλύτερο και περισσότερο διάλογο, το είπαμε από την αρχή, το ζητούμε ε, και από την Ευρώπη και από τις περιφέρειες και από τις διαχειριστικές αρχές και από τις εθνικές αρχές. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε καλύτερη πολιτική και μεγαλύτερο επίπεδο ε, ε, ιδιοκτησίας. Ε, ζητούμε επίσης μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε οι πολιτικές να είναι πιο καλά στοχευμένες. Ζητούμε ευκολότερο συντονισμό των ταμείων και των πόρων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι διαχειριστικές αρχές να συντονίζονται μεταξύ τους, γιατί διαφορετικά τίποτα δεν θα λειτουργήσει και σε πολλές ε, ε, περιπτώσεις ξέρουμε και σε πολλές ε, πόλεις ξέρουμε ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Επίσης χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία επιτόπου και επίσης καλύτερη καινοτομία, αστική καινοτομία που θα φέρει καλύτερη διακυβέρνηση. Έχετε ήδη από τον προηγούμενο Ιούνιο το έγγραφο που αφορά την πολιτική μας. Βεβαίως θέλουμε να διατηρήσουμε ισχυρή πολιτική και στρατηγική σε ολόκληρη την ε, Ευρώπη. Θέλουμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ε, και εταιρική σχέση η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Θέλουμε ε, ενδυνάμωση της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Θέλουμε ευελιξία και απλούστευση. Αυτή είναι η δέσμη την οποία ζητούμε. Δεν θέλω να επαναληφθώ γιατί ε, ούτως ή άλλως το έχετε λάβει το έγγραφο. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας λέει πώς είναι δυνατόν ε, ε, να επιβάλλεται. Δεν υπάρχει τρόπος, υπάρχει μόνο δυνατότητα μέσω ενός κώδικα δεοντολογίας. Θα πρέπει οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές ή οι κεντρικές εθνικές αρχές να λειτουργήσουν το πράγμα αυτό έτσι ώστε να λειτουργήσει καλά και να έχει αποτέλεσμα. Είπαμε ότι θέλουμε πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ των πόλεων, θέλουμε ε, στρατηγικό ευέλικτο πλαίσιο, ε, θέλουμε να δούμε κάποιες ε, περιφέρειες οι οποίες μπορεί να χρειάζονται κάτι παραπάνω από την πρόθεση της έρευνας και της ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι πολλά ζητήματα σχετίζονται και με τον έλεγχο και με τον λογιστικό έλεγχο και με τις ε, με, τις, ε, με τα κρατικά ε, συστήματα βοήθειας και οπωσδήποτε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το θέμα της ένταξης, της ολοκλήρωσης και μιλάμε για μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να είναι ισχυρή, η οποία θα πρέπει να ξεκινάει από πάνω και να πηγαίνει προς τα κάτω. Είναι σημαντικό λοιπόν να, το, να πιέσουμε διαδικασία προς αυτήν την διαδικασία. Επίσης, ε, καινοτομία. Η αστική καινοτομία αυτή τη στιγμή και οι δράσεις της είναι ε, ε, τυποτένιες. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Τώρα, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι πολύ ελέφαντας στο δωμάτιο σήμερα είναι η διασύνδεση ανάμεσα στην, πολιτική συνοχή και τις διαρθωτικές ε, ε, μεταρρυθμίσεις. Η πολιτική συνοχή όμως δεν μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο έτσι ώστε να ε, βγουν από το εθνικό επίπεδο αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Ούτως ή άλλως οι συστάσεις αυτές αναφέρονται στο πλαίσιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διασύνδεση να γίνει ε, με στή νοήματος, δηλαδή να υπάρξει διασύνδεση αλλά ε, όχι όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, με τρόπο αμφισβητήσιμο δηλαδή, αλλά με έναν τρόπο λειτουργικό και σωστό. Τέλος, ο ορισμός των ε, διαρθρωτικών ε, ε, μεταρρυθμίσεων δεν είναι κάτι απλό. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι η συγκρισιμότητα, η μετρησιμότητα κτλ. που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συνδυάσει κανείς. Όπως είπε όμως και ο Νικόλ Μικέλης και όπως μας κάλεσε να κάνουμε ο Νικόλα Ντε Μικέλης, ε, ε, ε, πρέπει να μπούμε στην συζήτηση αυτή. Εάν είναι κανείς στην συζήτηση, όπως οι πόλεις είναι έτοιμες να μπουν στη συζήτηση αυτή, θα πρέπει να αναλάβουν και περισσότερες ευθύνες οι πόλεις είναι διατεθειμένες να αναλάβουν ευθύνες, ε, να δουν με ποιο τρόπο οι μεταρρυθμίσεις μπορούν ε, να ενισχύσουν ε, κάποιες εκφάνσεις της τοπικής διακυβέρνησης. Η διασύνδεση ανάμεσα ε, στις αστικές και ε, μη αστικές περιοχές, περιοχές της ε, υπαίθρου. Επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι μια λειτουργική περιφέρεια, δηλαδή ένα λειτουργικό πεδίο το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από λειτουργικές μικρές περιοχές που μπορεί να είναι η γειτονιά μέχρι τη διεύρυνση της λειτουργικής περιφέρειας που μπορεί να είναι μια μεγάλη διοικητική περιφέρεια. Ε, θα πρέπει να αναπτυχθούν τοπικές πολιτικές, αλλά πάντα σε διάλογο με τις ομάδες ε, των ε, πολιτών. Θα πρέπει να διευρυνθεί αυτή η η διαδικασία η οποία θα πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω και που θα πρέπει να εμπλέκει τους πολίτες. Εάν έχουμε καλύτερη ιδιοκτησία σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, τότε θα είναι πιο αποτελεσματική και η συνολική πολιτική. Εν συμπεράσματι, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε συγκολητική ουσία για την Ευρώπη και αυτή η συγκολητική ουσία είναι η πολιτική συνοχή. Βέβαια, ξέρετε ότι οι συγκολητικέ ουσίε, αυτέ οι κόλλε, ε, μπορεί να κολλάνε στα δάχτυλα καμιά φορά. Επομένως ε, θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ουσία, το κατάλληλο υλικό, ε, το οποίο θα το δουλέψουμε σωστά για να έχει το σωστό αποτέλεσμα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση και αν ενεργήσουμε με τον τρόπο που ανέφερα προηγουμένως, η πολιτική συνοχής μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική συγκολητική ουσία που θα βοηθήσει το μέλλον της Ευρώπης. Το Reflection Paper ε, αναφέρεται μονάχα σε ένα σενάριο πολιτικής συνοχής. Αυτό δεν είναι σωστό. Ε, είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλοι ότι η πολιτική συνοχή ε, μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο για πραγματικά καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση και για το έγγραφο που έχετε διαμοιράσει προς τα μέλη μας. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Φαντεχίκ Βαλιέ, Γενικός Γραμματέας του CEMR, Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Εφόσον μου δίνεται η δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο λίγες μέρες μετά την ε, συνεδρίαση των ε, Γενικών Διευθυντών που αφορούσε το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να αναδείξω ε, τη διάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ευρώπη κρίνεται από τους πολίτες με βάση τα αποτελέσματα που προσφέρει. Πώς ανταποκρίνεται λοιπόν στα σημερινά προβλήματα και προκλήσεις ε, και πώς ε, προβλέπει και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Πώς ε, θα σταθούμε στο ύψος της ψηφιακής πρόκλησης. Τι μέτρα θα προτείνει για την απασχόληση των νέων που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, να μείνουν στις περιοχές και στις πόλεις τους και στις χώρες εννοείται. Τι μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την, ε, την μαζική εγκατάλειψη ορισμένων περιφερειών και άλλα ερωτήματα που ε, τίθενται και σε εσάς, φαντάζομαι, όταν πηγαίνετε στις εκάστοτε περιφερειές σας. Είμαστε Μέλλον, λοιπόν, είστε μάλλον εσεί ε, μέλη τη Επιτροπή ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη και ξέρετε ότι οι πόλει και οι περιφέρειε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά αυτέ τι προκλήσει. Χρειαζόμαστε επενδύσει. Το σχέδιο Juncker κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο στόχο είναι ε, να φέρει επενδύσει στον τομέα των υποδομών με μια πολιτική συνοχή και όλα αυτά πρέπει να πάνε ακόμα παραπέρα. Οι εκπρόσωποι τη τοπική αυτοδιοίκηση είναι πεπισμένοι ότι απαιτείται και απαιτούνται δημόσιε επενδύσει σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αποδίδει σημαντική σημασία στην ε, πολιτική συνοχής. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσει, καινοτομία, αλληλεγγύη και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επικρατείων της. Σκοπός ε, με αυτός είναι ο σκοπός με βάση ε, τη, των, τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές είναι και οι επιθυμίες των Ευρωπαϊκών πολιτών. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τέσσερα στοιχεία σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της πολιτικής συνοχής. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα κοινή στρατηγική μετά το 2020 βάσει ε, των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, πρέπει να βρούμε στόχους για το 2030 αλλά και με βάση και ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του, 2000, του ΟΗΕ, το θεματολόγιο 2030, την ε, κλιματική συμφωνία των Παρισίων. Αυτό θα μας δώσει έναν στατηγικό προσανατολισμό ε, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και θα μας επιτρέψει να ταλοποιήσουμε όλα αυτά καλύτερα σε όλη την Ευρώπη. Η πολιτική συνοχή σε αυτή την πραγματική περίοδο έχει υιοθετήσει μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ ε, κυβερνήσεων και διαφόρων φορέων. Πρέπει λοιπόν να υποπτεύσουμε αυτή την, πλήρη ε, υλοποίηση αυτής της πολιτικής και αυτό εξαρτάται από την καλή συνεργασία μεταξύ δήμων, ε, πόλεων, περιφερειών. Η μελλοντική πολιτική συνοχή θα πρέπει να εμπλέξει σε μεγαλύτερο βαθμό την, το τοπικό επίπεδο όχι μόνο για τη διαβούλευση και επιλογή έργων, αλλά και για την ιεράρχηση επενδυτικών προτεραιοτήτων. Υπάρχει κώδικα διοντολογία σε ό,τι αφορά τι αρχέ των εταιρικών σχέσεων. Θα πρέπει να αποτελέσει δεσμευτικό στοιχείο οποιασδήποτε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση. Ε, και σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την ενίσχυση ε, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ε, ζητούμε να συμμετάσχουν ε, και οι αρχές αυτές λοιπόν. Τρίτον, θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εδαφική διάσταση για να ενισχύσουμε την ολοκληρωμένη υλοποίηση της πολιτικής. Πρέπει λοιπόν και οι πόλεις και οι ύπεθρος να αναπτυχθούν από κοινού σε όλη την Ευρώπη πόλεις ε, και χωριά καταλαβαίνουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για την ε, υλοποίηση δράσεων προκειμένου να αναπτυχθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και εμείς έχουμε ένα μότο που λέει ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ε, εδαφική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν οι σχετικές στρατηγικές, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ολοκληρωμένες τέτοιες στρατηγικές. Σκοπός είναι να ενθαρρύνουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα καλύπτει συγκεκριμένε ανάγκες της κάθε ζώνης. Θέλουμε να διευρύνουμε τα κριτήρια κατανομής πόρων μεταξύ των επιμέρους ε, περιφερειών, πέρα του ε, ΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. και έτσι θα έχουν και τους κατάλληλους πόρους ε, οι περιφέρειες. Μετά, όπως ε, αναφέρεται και στην τελευταία έκθεση για τη συνοχή, πρέπει να συγκεντρώσουμε ε, τα κονδύλια για τους διαχειριστές και τους δικαιούχους. Πρέπει να θεσπίσουμε ένα κοινό σύνολο κανόνων για όλα τα ταμεία για να διευκολύνουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Χρειαζόμαστε επίση μεγαλύτερη ευελιξία, όπω ανέφερε η Αναλύζα προηγουμένω. με λιγότερε προκαθορισμένε ε, κατανομές και κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσων υλοποιούν την πολιτική. Αυτό θα επιτρέψει τη διαδικασία και την απλούστευσή τη, ιδίως ό,τι φορά του ελέγχου και τις επιθεωρήσεις και θα επιτρέψει στους Δήμους και στους ε, δικαιούχους με λιγότερη εμπειρία να συμμετάσχουν ε, και να εμπλακούν στην πολιτική η πολιτική συνοχή είναι αυτή που βρίσκεται υπό πιο στενό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο ε, παρακολούθησης με ένα πολύ μικρό περιθώριο σφάλματος, μόλις 5%. Και σε ό,τι αφορά και την αρεσιμότητα, που είναι κάτι που αναφέρθηκε προηγουμένως, η μεταβλητή προσαρμογή δεν μπορεί να είναι πολιτική συνοχή. Υπάρχουν και άλλε ευρωπαϊκέ πολιτικέ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικεντρωθούμε στι ε, κοινέ μα αξίε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να στερούμε ε, από τις ε, περιφέρειες τις ευκαιρίε να αναπτυχθούν και να υποστηρίξουν τους πολίτες τους. Εμείς ε, είμαστε πλήρως διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το πράττουμε για να αναπτύξουμε μια πιο ισχυρή ε, πολιτική συνοχή μετά το 2020. Με την στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο, τον επόμενο Σεπτέμβριο θα προγραμματίσουμε μία σειρά τέτοιων συζητήσεων σε 8 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων Αυστρία, Βέλγιο, Σουηδία, κάτω και Ιταλία, ε, για να αναδείξουμε την προσταθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής ε, για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος. Υπάρχει και ένα βιβλίο που έχουμε εκδώσει, Ευρώπη 2030, μετά από δύο έτη στοχασμού και συζητήσεων με, τις, ε, με πολίτες, με αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, είχαμε παρεμβάσεις από πάνω από 100 ε, τοπικούς εκπροσώπους από όλη την Ευρώπη και σας ε, προσκαλώ και στη διάσκεψή μας για την ε, ισότητα, την ποικιλομορφία και την συμπερίληψη που θα γίνει τον Ιούνιο 11 έως 13 Ιουνίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και χαίρομαι που μπορέσαμε να το δούμε και για την πρόσκληση ευχαριστούμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακολουθήσουμε τη διαδικασία στους διάφορους οργανισμούς. Και τώρα η κυρία Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέας της Διάσκεψης των Περιφερειακών Θαλασσίων Περιοχών Απόψεων που θα κάνουμε για την έκθεσή σας κύριε Ζουλό. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Εμείς ως οργανισμός πάντα προσπαθούσαμε να βρίσκουμε λύσεις σε δύσκολα θέματα με προτάσεις και να ε, γνωρίζουμε όλοι σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020 ξέρουμε ότι θα πληγεί από περικοπές η πολιτική συνοχής. Επίσης ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα περιλάβει το κοινωνικό ταμείο. Το θα ενισχυθεί. Ξέρουμε ότι οι εξάντε ερεσιμότητες θα παραμείνουν και ξέρουμε ότι οι μακροοικονομικές ερεσιμότητες θα υπάρχουν. Δεν θα βγουν από την εικόνα παρά τη θέληση και επιθυμία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάει να εντάξει κάποια κίνητρα για να συνδέσει την πολιτική, συνοχή για να υποστηριχθούν στα κράτη-μέλη διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να γνωρίσουμε γιατί αυτά ε, δίνουν το πλαίσιο. Ο κ. Δεμικέλης μας έδωσε το πλαίσιο ότι δεν τέλειωσε η διαδικασία και τώρα κορυφώνονται οι δύσκολε διαπραγματεύσει όταν δηλαδή και είναι έγκαιροι η συζήτηση που κάνουμε με κάποιες προτάσεις μας που υποβάλλουμε και σε εσά και στην Επιτροπή Ρέτζη και στην Επιτροπή. Να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό αρχικά. Ακούσαμε μέχρι τώρα και ο κύριος Έτιγκερ ήταν ξεκάθαρος ότι θα έχουμε μία τρύπα, είπε, λόγω του Brexit, την έξω. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα, δεν μπορούμε να το ε, παραμελήσουμε. Το άλλο είναι και πολλοί επίτροποι και ο Έτιγκερ και ο Γιούγκαρ και άλλοι το συζητούν γιατί είναι στο χέρι τους αυτό στα πλαίσια του ΠΔΠ πρέπει να δούμε νέες προτεραιότητες εδώ και τις τωρινές η πολιτική συνοχή ε, είναι παραδοσιακή με την πολιτική πρέπει να πούμε ότι κάποιες ε, τωρινές ε, προτεραιότητες δεν είναι ξεπερασμένες, υπάρχουν εδώ και 40 χρόνια, έδωσαν αποτελέσματα που τα είδαμε και στην έκθεση για τη συνοχή και σε άλλα έγγραφα προβληματισμού της συνοχής όταν μιλάγαμε για το μέλλον της Ευρώπης. Έδειξαν όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι θεμελιώδες. Δεν μπορεί να έχεις ε, μαζεράτη, λάμπερτ ε, με δύο ρόδες μόνο και να λείπουν δύο τέτοιο αυτοκίνητο δεν φτιάχνουν δρόμους υπερηφέρειε και κτίρια, αλλά για να γεφυρωθεί το κενό. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτή είναι μια τωρινή, παραδοσιακή και μελλοντική. Ποτέ δεν είχε ακουστεί η πιθανή αύξηση. Ο κύριος Έτιγκερ μιλάει για 1,15 ή 1, κάτι. Και είπα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή τι σημαίνει αυτό. Πάμε τώρα στην καθαυτό πολιτική συνοχή πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την πολιτική συνοχή αφού τελειώσουμε με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και πώς μπορούμε να εντάξουμε τις, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ε, στην εισαγωγή αυτά τα πράγματα υπάρχουν, δεν είναι καινούρια, υπάρχει σύνδεση. Υπάρχουν διάφορα άρθρα στην, στον κανονισμό. Υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη ήδη να κατανείμουν χρήματα από τη συνοχή για να κάνουν μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια του εξαμήνου. ε, ε αφαιρεθεί ο λόγος ύπαρξης της πολιτικής. Είναι σημαντικό, αφού λοιπόν, όπως είπαμε, δεν υπάρχει συνολική στρατηγική για να δούμε πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα... Λοιπόν, εμείς οι ίδιοι να θέσουμε στόχους ε, που να ισχύουν πάντοτε. Και όταν υπάρχουν συζητήσεις και επικίνδυνες προτάσεις, όπως η πιλωτική πρόταση από την ε, μεταρρύθμιση της ΟΝΕ που είπαν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια μεταρρυθμίσεις. Δεν ε, είμαι κατά των ε, μεταρρυθμίσεων και να υπάρχει δυναμική για να υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά πώς θα εξηγήσουμε ότι θα πληρώσουμε τα κράτη-μέλη από τον ενωσιακό Προϋπολογισμό για να τα κάνουν αυτά. Γιατί αν είναι αναγκαίε οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να τις κάνουν ούτω ή και προς ποια κατεύθυνση. Έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα σας το στείλουμε σήμερα το απόγευμα σε όλους σας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να, δούμε, να σας δείξουμε τι πιστεύουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε μια σύνδεση. Έχουμε ε, λεπτομέρειες που είπες Λάμπερτ και θα τις λάβεις. Και η πολιτική. Μην εργαλειοποιούμε την πολιτική. Το Εύση, το, το, για τις στρατηγικές επενδύσεις, μάλιστα, είναι εργαλείο, είναι ένα μέσο, αλλά η πολιτική είναι πολιτική, η διαφορά είναι μεγάλη. Ε, λοιπόν, δεν είναι μόνο η σύνδεση. Το ερώτημα είναι τι σύνδεση θα είναι αυτή. Τι θέλουμε να... Ε, δεν, ε, το, το, το, το, δεν έχουμε τη στρατηγική που χρειαζόμαστε για να δούμε ακριβώς ε, ποιοι είναι οι στόχοι της πολιτικής συνοχής, οπότε είναι δικό μας θέμα να τους ορίσουμε, όπως είπε και ο κύριος ε, Ντεμικέλης, στόχοι σε περιφερειακό επίπεδο, να δούμε εφαρμοστούν μακροπρόθεσμα από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Ένα άλλο που πρέπει να γίνει τώρα, νομίζω ότι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, είπε ότι ιδιωτικό τομέα, ε, κοινωνικο-οικονομική εταίρη, θα ήθελα να σας καλέσω και να συνδιοργανώσουμε, κυρία Πρόεδρε, θα θέλαμε μια συνάντηση στη Γαλλία, η Τοσκάνη, στην... Ε, και μία στη Γερμανία για να φέρουμε τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους και τους δικαιούχους και ε, για να αποδείξουμε ότι η πολιτική αυτή έδωσε στους δικαιούχους ε, αποτελέσματα. Τα χρήματα φεύγουν από τα κανείς, δεν τα παίρνει πίσω. Ε, οπότε δεν μπορούν καμιά φορά όταν, έχουμε αυτούς που, όταν κάνουμε τη συζήτηση για αυτούς που πληρώνουν και γιατί να αυξήσουμε τον προπολογισμό ε, αυτό εξηγεί. Και φαίνεται ότι στην πράξη υπάρχουν παραποτελέσματα που μένουν στις τσέπες των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ε, και είμαι σίγουρη ότι και εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι συνάδελφοι θα θέλουν να συμμετάσχουν. Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε τη θέση σας. Θα μας τη στείλετε σήμερα. Οποιαδήποτε προσπάθεια, οποιαδήποτε συζήτηση μπορεί να βοηθήσει το, στη συνολική συζήτηση συνοχής, χωρίς όμως αναφορά στο κοινωνικό ταμείο που ε, είναι τμήμα σημαντικό ε, της ε, πολιτικής συνοχής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας να διατηρήσουμε το οικοδόμημα ενωμένο, να βλέπουμε τους στόχους, να ο οποίο είναι γενικό Γραμματέας ε, της ε, των συνοχή, Συνοχής. Ε, μιλάω τελευταίος και ίσως θα πω δύο-τρία πραγματάκια που να τα έχετε ήδη ακούσει. Δεν υπάρχει ε, σημαντικότερη πολιτική για την ε, ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική ε, σύγκληση από την ΕΣΕ. Έχει υποστηρίξει τις περιφέρειες, την δημιουργία θέσεων εργασίας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στην τελευταία προγραμματική περίοδο δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας και εκατομμύρια παιδιά ότι ε, υπάρχει γενικά μια απογοήτευση και απομάκρυνση από την Ευρώπη, πιστεύουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την πολιτική συνοχή έτσι ώστε να ε, κάνουμε πιο θελκτική την Ευρώπη. Να μην λησμονούμε όμως τη γενικότερη εικόνα πέρα από τα οποιαδήποτε μέρους προβλήματα και έστω και αν εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλήσει και διαφορέ, όπω αναφέρθηκε και προηγουμένω, εξακολουθεί η πολιτική συνοχή να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Θα πρέπει γρήγορα ε, σε ευφυείς ε, καινοτόμες ε, επενδύσεις ε, οι οποίες θα είναι αντίστοιχες της νέας ε, η διαδικασία των building blocks για την ε, πολιτική συνοχή και από τότε έλα εδώ να σας παραπέμψω στο έγγραφο εργασίας μας. Πρώτον θέλουμε απλουστευμένες διαδικασίες, ευκολότερες διαδικασίες και κακού ελέγχου που βασίζονται στις επιδόσεις είναι ένα σημαντικό έργο εργαλείο. Επίσης, ε, μείωση των ε, ε, μεγαλύτερη ευελιξία έτσι ώστε να προτείνουμε λύσεις πιο συγκεκριμένες και προσανατολισμένες προς ειδικέ καταστάσεις. Συνοχή, επομένως, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική συνοχής που θα λαμβάνει υπόψη τοπικό, περιφερειακό κλπ. Αυτό αυτός που σας ανέφερα είναι ένας κατάλογος επί των οποίων έχουν συμφωνήσει τα μέλη μας ε, και ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κινούνται οι διαδικασίες εντός αυτών των, των πεδίων προτεραιότητας. Η εδαφική συνεργασία είναι πάρα πολύ ε, για την προώθηση των ανταλλαγών εμπειριών και βελτίστων πρακτικών. Ε, οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να πάρει κονδύλια από τους στόχους της ε, πολιτικής ε, συνοχής δεν βρίσκουν τις περιφέρειες σύμφωνες. Να γίνει ένα είδος καρότου και μαστιγίου που θα χρησιμοποιείται αναπερίπτωση. Θέλουμε να χρησιμοποιούνται και να δαπανούνται σωστά και αποτελεσματικά τα κονδύλια της πολιτικής ε, ε, Το τελευταίο καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πιστεύουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ε, εργαλεία αυτά Μονάχα όμως εάν ε, συμπεριληφθούν στις διαδικασίες ε, και οι τοπικές περιφερειακές αρχές ε, θα καλυφθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες των πολιτών σε περιφερειακό επίπεδο από την πλευρά των περιφερειών με τρόπο διαρθρωμένο και με τρόπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η λογοδοσία καθώς επίσης και ε, η ιδιοκτησία. Ε, το επόμενο πολιτές σε τις πολιτικές οι οποίες μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία ε, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και την αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Τούτων ελεχθέντων πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας, ε, ε, ε, ένας κρίκος ο οποίος λείπει να δουλέψουμε όλοι μαζί εμείς τις συμμαχίες για την πολιτική συνοχή. Αναμφιβόλως οι πόλεις και θα δουλέψουν και θα δώσουν τον αγώνα μαζί μας. Thank ο Σέτιγκερ δήλωσε τα εξή. Η κοινή γεωργική πολιτική, η πολιτική συνοχή και η έρευνα θα παραμείνουν στο επίκεντρο ε, των προτεραιοτήτων του προπολογισμού για την επόμενη δεκαετία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Δύο ερωτήσεις. Αφενός, για την Συμμαχία Συνοχής. Την πρωτεύουσα. Πραγματικά είναι από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Γιατί βλέπουμε και στο Twitter ε, με το hashtag Cohesion Έχουμε τους ηγέτες και τους ουραγούς. Αυτό συνδέεται και με την έρευνα, τον ανταγωνισμό. Πείτε μου λοιπόν δύο πράγματα για την ευφύ εξειδίκευση και την επόμενη φάση αυτού του χειρήματος. Μίλησα προηγουμένως για τη Μαζεράτη, γιατί νομίζω ότι η ευρωπαϊκή οριζόντια πολιτική κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το μια Μαζεράτη, ένα Airbus. Ακόμα και ο ΣΑ λέει ότι οι πολιτικές μας είναι σωστές. Έχω και εδώ ένα άρθρο που λέει ότι η Ευρώπη είναι σαν ένα Airbus που προσπαθεί να προσγειωθεί χωρίς όμως τον κατάλληλο εξοπλισμό. Όπως των διαφόρων οργανώσεων για τα όσα είπαν και γιατί στην ουσία υποστηρίζουν ε, την ε, ε, πολιτική Συνοχή, ε, ε, άλλωστε το έλεγε και ο συνάδελφο, δεν είχαμε καμία αμφιβολία, το είπε και ο συνάδελφο ότι όλοι είμαστε μέλη αυτού του, αυτού του συνάδελφου, οποία πιστεύω ότι αναδύθηκαν ε, και από τα δύο πάνελ, του δύο γύρου ε, συζήτηση. Το πρώτον, ότι θα πρέπει να παραμείνει πολιτική για όλε τι περιφέρειε, αλλά θα πρέπει να έχει και την δυνατότητα στο εσωτερικό των περιφερειών και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τη κάθε περιφέρεια. 2030 όμω εντό τη στρατηγική αυτή πιστεύω πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε ε, αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Δηλαδή να βοηθήσουμε τις περιφέρειες που μένουν πίσω, ε, να βοηθήσουμε αυτές τις περιφέρειες ε, που αντιμετωπίζουν το καινούριο πρόβλημα να έχουν παγιδευτεί στο μέσο εισόδημα. Δούμε και τα προβλήματα των περιφερειών που έχουν χαμηλή δημογραφική πυκνότητα. Ε, ε, λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να διορθωθούν σωστά οι προτάσεις για το 2030. Το επόμενο είναι να μην τα φορτώσουμε όλα στην πολιτική συνοχή. Είναι γεγονό ότι θα πρέπει να τη ε, σε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά ε, του διαγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπούντα. Ε, που είναι και τα ίδια πολιτικά κόμματα καμιά φορά με του Πρωθυπουργού κλπ. Καμιά φορά δημιουργείται μια δυναμική ανθρώπων που θέλουν να ακούσουν και θέλουν να δουν γιατί τα αποτελέσματα που έρχονται σε, σε αυτούς ε, υλοποιούνται αλλά πολλέ φορέ ο υπουργό ε, δεν ε, έχει ενημερωθεί, ενώ υπάρχουν δραστηριότητε. Και με κράτο μέλος και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μπορεί να είναι σε επίπεδο γενική διεύθυνση ή σε επίπεδο κρέτσου. Πάντως θα υπάρχει κάποιος ε, από εκεί για να γίνει συζήτηση με αυτούς που πληρώνουν στον προϋπολογισμό. Για τις συνεισφορές των κρατών μελών, το είπε Έτιγκερ. Οπότε και ό, από ό,τι είπε και Ντεμικέλης, αν έχουμε λιγότερα χρήματα θα επικεντρωθούμε περισσότερο. Η έξυπνη εξειδίκευση των πόλεων, ε, θα έλεγα και οι έξυπνες πόλεις, ε, απαιτούν μια εξυπνή σε θεματικά θέματα, σε κάποιες προτεραιότητες που είναι σημαντικές. Οι συνέργειες με τα ταμεία δεν είναι εύκολες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε συνέργειες με τα ταμεία, αλλά είναι τόσο διαφορετικοί οι κανόνες που ισχύουν. Εγώ θα ήμουν ευτυχής να έχω συνέργεια μεταξύ του Ταμείου συνοχή για την καινοτομία και το πρόγραμμα έρευνας, αλλά δεν είναι εύκολο. Και αυτή δεν είναι πολύ έξυπνη, έχει δυσκολίες. Αν γίνει απλοποίηση με τρόπο ώστε να αλλάξουν όλα αυτά ριζικά και να βοηθηθούν οι δικαιούχοι να φροντίσουν ότι οι κανόνες τους εξυπηρετούν, ε, εντάξει, αλλά δεν νομίζω να γίνει αυτό για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και τέλος, δεν το είπαμε, αλλά είναι θεία άμεσα η πρόταση από εσάς η Βουλγαρική Προεδρία είπε ότι θα το πιέσουν να γίνει συνάντηση και να συνεννοηθούν και με την Αυστριακή Προεδρία για να τελειώσουμε στα πλαίσια αυτής της θητείας του Κοινοβουλίου. Ελπίζω αλλιώς θα γίνονται καθυστερήσεις η μία μετά την άλλη. Ε, δεν το αναφέραμε αυτό, αλλά μου φαίνεται και αυτό είναι σημαντικό, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή. Ευχαριστώ, Φρέντερικ. Ευχαριστώ. Λίγα σχόλια. Δεν θα επαναλάβω αυτό που είπε η συνάδελφος Ελένη. Για να απαντήσω ε, σε αυτό που είπατε για τον κύριο Έτιγκερ και τα ίδια ακούω παντού όπου πάω, όλοι ε, μιλούν για την πολιτική του θεμελιώδους πυλώνα, αλλά πρέπει να ξανασκεφτούν τον προϋπολογισμό, γιατί υπάρχουν και άλλες πολιτικές που πρέπει να υποστηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν φοβόμαστε τόσο ότι θα ε, εξαφανιστεί η πολιτική συνοχής και στο Συμβούλιο ε, θα πούνε ότι ναι, πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά το θέμα είναι τι θα μείνει, πόσο θα την στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο διατεθειμένα είναι τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν στις διαθωτικές αλλαγές και την πολιτική συνοχής και στα διαρθρωτικά ταμεία, συγγνώμη. Και αυτό θα το παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά. Να, μάλλον, να επιμείνω στη σημασία της σχέσης ε, μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών. Θα πρέπει να επιμείνουμε να ζητήσουμε από τις περιφέρειες ε, να δημιουργήσουν την ικανότητα για τέτοιες συμπράξεις. Δεν θα αναπτυχθούν οι Μητροπόλεις αν η ενδοχώρα ε, διψάει για ανάπτυξη. Επίσης υπάρχει ανάγκη να μην δημιουργήσουμε ένα συγκεντρωτικό σύστημα παροχής της πολιτικής συνοχής ε, οι Γάλλοι ξέρω ότι αρέσκονται στην ε, συγκεντρωποίηση, σε ένα συγκεντρωτισμό, αλλά είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για διάλογο ε, στα πλαίσια συμπράξεων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών αρχών και κυβερνήσεων. Για τη συμμαχία να πω ότι αυτό που κάνουμε με τους περιφερειακούς ε, διαλόγους που οργανώνουμε Στι 8 χώρε που συνεισφέρουν στον προπολογισμό είναι ένα τρόπο να εντάξουμε κι άλλου ε, εμπλεκόμενου ε, και τα περισσότερα μέλη μας, οι Εθνικέ Ενώσεις Δήμων και Περιφερειών, ήδη είναι μέλη στη Συμμαχία. Ελπίζω ότι όλοι θα είναι και βέβαια θα εργαστούμε όχι μόνο με τους συνήθεις υπόπτους και τους υποστηριχτές της Συμμαχίας, αλλά θέλουμε να φτάσουμε σε εκείνους που ωφελούνται από την πολιτική συνοχή και καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουν κιόλας ότι ωφελούνται. Ε, μετά το Brexit θυμάμαι ότι το Euronews είχαν πάρει συνέντευξη από έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο από την Κορνουάλη και έλεγε «Εγώ δεν το κατάλαβα ότι δεν θα παίρνουμε λεφτά μετά τον Brexit από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ψήφισε τον Brexit και μετά κατάλαβε ότι η περιφερειακή πολιτική στήριζε αυτά που έκανε αυτό στο Δήμο του. Λοιπόν, ε, και αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτή είναι, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ναι, οι ε, που εκπροσωπούμε είναι ο χώρος όπου είναι αν θέλετε το σημείο σύνδεσης, μια παραμεθόρια άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Και εμείς διοχετεύουμε το μήνυμα τους τώρα γιατί σύνδεση μεταξύ ταμείων θα τα αξιοποιήσουν. Αυτό είναι κομμάτι μιας δουλειάς που δεν θα έπρεπε όμως να κάνουμε πια γιατί είναι πάρα πολύ χρονοβόρος και εν... καλό είναι αυτό να γίνεται. Τώρα, για την ε, Συμμαχία Συνοχής, το γεγονός ότι υπάρχει Συμμαχία Συνοχής είναι πράγμα καλό. εξειδίκευση. Εδώ πρέπει να μιλάμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα, πρέπει να μιλάμε για την αστική ανάπτυξη και εκεί το, το κοινωνικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πόλεις έχουν όλο και περισσότερο σημαντικά στοιχεία τους καθαρούς ε, ε, συμβάλλοντες της πλούσιας χώρες, οι οποίες ε, δεν θέλουν πολλές αλλαγές. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε να